Uh, Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε χωρίς να εξαντλήσουμε το ακαδημαϊκό τέταρτο. Έχω τη χαρά και την τιμή να προεδρεύω στις απογευματινές μας εργασίες, τουλάχιστον στο πρώτο γύρο με θέμα τις οικονομικές προκλήσεις, ανάπτυξη, συνεργασία και κρίση. Και το επαναλαμβάνει και στα αγγλικά η πρόεδρος. Επειδή δεν θέλω να κόψω χρόνο από τους καλεσμένους ε, ή από το ακρατήριο. Θα είμαι εξαιρετικά λακωνική και θα συνοψίσω την ομιλία μου σε δύο σημεία, τα πιο βασικά. Το πρώτο αφορά το πώς είναι εξουσίες, το κοινοβούλιο, οι κυβερνήσεις, οι πολιτικοί ηγέτες αντιμετωπίζουν τις ε, σημερινές ε, οικονομικές και άλλες προκλήσεις. Η χειρότερη είναι η ανεργία των νέων, που ταλάνιζε την κοινωνία και στο προηγούμενο καθεστώς, αλλά με τις επαναστάσεις δημιουργήθηκε η ελπίδα και η προσδοκία στους νέους ότι θα υπάρξει μια γρήγορη βελτίωση, κάτι που δεν έχει συμβεί. Οπότε πώς θα διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι σε πολλά Ισλαμιστικά κόμματα διαφαίνεται η επιθυμία της αρχής των αρχών, των Ισλαμικών αρχών για την οικονομία, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν τέτοιες Ισλαμιστικές αρχές για την οικονομία, η Ισλαμιστική προσέγγιση της οικονομίας. Το θέμα είναι πώς βλέπετε ε, τις προκλήσεις ε, υπό το πρίσμα αυτών των Ισλαμιστικών οικονομικών αρχών και πώς, θεωρεί, πώς μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι οικονομίες που θα διέπονται από τέτοιες Ισλαμιστικές οικονομικές αρχές ε, θα μπορέσουν να ενταχθούν σε ένα παγκόσμιο σύστημα που σίγουρα δεν είναι συνεκτικό, αλλά σε μεγάλο βαθμό κυριαρχείται από τους κανόνες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Η Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου δεν είναι ένα άναρχο όργανο. Αντίθετα, είναι ένα όργανο, μια οργάνωση από την οποία εκπορεύονται ε, πολύ και αυστηροί μερικές φορές εμπορικοί κανόνες. Έχουμε πολλούς ε, δεκεκριμένους καλεσμένους. Θα σας τους παρουσιάσω πρώτα και μετά θα τους δώσουμε το λόγο. Πρώτη καλεσμένη συγγετριά μας, η κυρία Σάρα Τσάιες, που ε, εκπροσωπεί το Ίδρυμα Κάρνεγκη, για τη διεθνή ειρήνη με έδρα τη Washington, αν δεν κάνω λάθος. Η κυρία Τσέις έχει ένα πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με τους συσχετισμούς μεταξύ της οξίας ε, ε, διαφθοράς στο δημόσιο τομέα και της έξαρσης ε, των εξτρεμιστικών κινημάτων. πολύ εντυπωσιακό. Ε, η κυρία Τσάγης έγραψε το βιβλίο «Τιμωρία της αρετής». Ε, ματιά του Αφγανιστάν υπό το Σταλιμπάν. Επίσης, ε, σύνταση άρθρα και σημαντικές εφημερίδες. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, να δώσω το λόγο στην κυρία Τσέιες ή μήπως κάνω λάθος. Α, όχι, εσύ θα μιλήσω στο τέλος. εντάξει, ωραία. Ας προχωρήσουμε τότε στους άλλους καλεσμένους μας. Πρώτα στον κύριο Σαμεχ Φωζή Χάινεν, που είναι από την Αίγυπτο, μέλος του Συμβουλίου Σούρα, Ο Δόκτωρ Φωζή ήταν και διευθυντής του Κέντρου ε, Αναπτυξιακών Σπουδών που λειτουργεί από το 2009 στην Αλεξάνδρεια και είναι και σύμβουλος ε, οικογενειακός ε, για διάφορες τοπικές και διεθνείς οργανώσεις όπως είναι η USAID και η UNESCO. Έχει δακτορικό στην δημιουργία του κοινωνικού κεφαλαίου και ένα μάστερ σε θέματα λογιστικής και διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Κάιρο. Και επίσης ε, έχει μεταπτυχιακό και από το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ. Και έχουμε και τον κύριο Μοχάντα Σαλέμ που είναι υπουργό Γεωργίας της Τινησίας και μέλος του κόμματος Ενάχντα Είστε λοιπόν υπουργό Γεωργία και ήσταν από τους ηγέτε του Κόμματο Ενάχτα και μέλος του εκτελεστικού γραφείου από το 1989. Είστε μάλιστα εμπειρογνώμων για τους ε, υδατινού πόρους, ε, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και καθηγητής στην Γεωργική Σχολή της Τινησίας. Επίσης, έχετε σπουδάσει και στην Ανώτατη Σχολή του Στρασβούργου και έχουμε και τον κύριο Χακίμα Φασιλή, μέλος του κόμματος ε, ε κυρία μάλιστα Φασίλη, συγγνώμη, μέλος του κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξης ε, και μάλιστα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο 2. Και ε, βουλευτής της Μαροκινής Βουλής και μέλος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, καθώς και καθηγήτρια στην νομική σχολή της Μαμέντια, που κάνετε μάθημα για τα μικροοικονομικά. Ε, δεν θα ενδώσω στο κλισέ οι κυρίες προηγούνται. Δεν θα δώσω πρώτα το λόγο σε μια κυρία. Με, με ενοχλούν τέτοια κλισέ. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Σαλέμ, τον Υπουργό Γεώργιας της Τινησίας, για να δώσει τον αρκτήριο λάκτισμα και για 10 λεπτά. شكرا بسم الله الرحمن Σας ευχαριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωκοινοβούλιο για την πρόσκληση αυτή που μου απέφθινε, γιατί θεωρούμε πως ε, υπάρχει ανάγκη για έναν ειλικρινή διάλογο ανάμεσα στις δύο όχθες της Μεσογείου. Συνήθως ακούτε άλλους να μιλούν για μας. Σήμερα όμως έχετε την ευκαιρία να μας ακούσετε άμεσα. Απ' την άλλη πλευρά, με χαρά άκουσα τα όσα υπόθηκαν σήμερα το πρωί, κυρίως από πλευράς του κυρίου Μπρόκ και του κυρίου Βημό και την... είδα ότι υπάρχει μεγάλη κατανόηση για τα όσα συμβαίνουν στην άλλη άκρη, στην άλλη όχθη της Μεσογείου. Εξακολουθούμε, δεν να αποκαλούμε την Αραβική Άνοιξη Άνοιξη και θα συνεχίσουμε να την αποκαλούμε Άνοιξη και στο μέλλον. Αν όμως ορισμένοι θέλουν ή επιμένουν για να την αποκαλούν ε, ε, Ισλαμικό χειμώνα, να θυμίσω ότι ακόμα και ο χειμώνας στις χώρες μας είναι ηλιόλουστος. Και έπειτα ο χειμώνας είναι ο μήνας ε, των βροχών και ως Υπουργός Γεωργίας θεωρώ τον χειμώνα ως την πιο όμορφη εποχή, γιατί χωρίς ε, το, τις βροχές η γεωργία δεν προοδεύει. Σήμερα λοιπόν ε, η σημερινή ομιλία θα αφιερωθεί στην οικονομία. Αλλά πριν να μιλήσω για το σήμερα να σας πω τι κληρονομήσαμε από το προηγούμενο καθεστώς. 800.000 άνεργοι, από τους οποίους 250.000 πτυχιούχοι με πανεπιστημιακά πτυχία. Αυτό κληρονομήσαμε από το καθεστώς του Μπεναλή. Επίσης, ανάπτυξη μείον 2,2. Και παρά τις πολυάριθμες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, ως κυβέρνηση καταφέραμε να βελτιώσουμε το ποσοστό ανάπτυξής μας και έχουμε φτάσει στο 3,6%. Εάν δεν συγκρίνουμε το ποσοστό αυτό με το ποσοστό των γειτόνων, είμαστε πολύ πάνω από τους γειτονές μας που δεν αντιμετωπίζουν δε, τα ίδια προβλήματα όπως εμείς ως ε, κληροδότημα του παρελθόντος. Ε, η επανάσταση είναι σαν τους σεισμούς. Έχουμε τον κύριο σεισμό και μετά τους μετασεισμούς που ακολουθούν τον κύριο σεισμό, την πρώτη δόνηση. Και μπορούμε να πούμε ότι οι μετασυσμοί είναι πολυάριθμοι. Όπως σας είπα, το ποσοστό ανάπτυξής μας είναι της τάξης του 3,6% αυτή τη στιγμή, αλλά στο επίπεδο της απασχόλησης καταφέραμε σύμφωνα με ανεξάρτητες εκτιμήσεις καταφέραμε να δημιουργήσουμε 112.000 θέσεις απασχόλησης. Αυτά τα νούμερα δε είναι από το περασμένο Δεκέμβριο. Πάνω από 20.000 θέσεις στο δημόσιο τομέα Αυτές οι θέσεις ε, δημιουργήθηκαν μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει δηλαδή σύνολο 338.000 θέσεις απασχόλησης. Εάν ε, συγκρίνουμε αυτά τα νούμερα με το τι είχε καταφέρει την νησιακή οικονομία πριν από την Επανάσταση, φέτος είναι η καλύτερη χρονιά για την, ε, την νησιακή οικονομία όσον αφορά την απασχόληση. Για το 2007 που ήταν η καλύτερη χρονιά του παλιού καθεστώτος είχαν δημιουργηθεί 7.000 θέσεις απασχόλησης. Δηλαδή εμείς καταφέραμε να δημιουργήσουμε σχεδόν το διπλάσιο θέσεων από ότι το παλιό καθεστώς μέσα σε δύο χρόνια. Όσον αφορά τώρα όσους ε, παραμένουν άνεργοι, 670.000 νέοι άνεργοι που δεν κατάφεραν να βρουν δουλειά, για εκείνους η κυβέρνησή μας έχει αποτύχει, γιατί μετά από δύο χρόνια μετά την Επανάσταση εξακολουθούν να περιμένουν να βρουν μια θέση. Και αυτό την ε, προσωπεύει βέβαια ε, πολύ σοβαρό ε, πρόβλημα. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα κόμμα ούτε στην αντιπολίτευση ούτε στην κυβέρνηση που να έχει υποσχεθεί να ε, φτιάξει τόσες ε, θέσεις απασχόλησης όσοι είναι οι άνεργοι. Πρέπει δηλαδή να διαρωτηθούμε πώς θα πείσουμε αυτούς τους νέους που δεν κατάφεραν να βρουν θέση ότι υπάρχουν ακόμα δυνατότητες, ότι η οικονομία μας βελτιώνεται και ότι στο μέλλον θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες. Το θέμα λοιπόν είναι πώς δεν καταφέραμε να κάνουμε καλύτερα ακόμα, να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Ξέρετε πως η παγκόσμια οικονομία ε, είναι αλληλένδετη. Εμείς είμαστε πολύ στενά συνδεμένοι με την ευρωπαϊκή οικονομία και δυστυχώς η κρίση που πλήττει την Ευρώπη οδήγησε στο ότι τα εργοστάσια στην νησία, ιδιαίτερα αυτά που ε, κάνουν υπεργολαβίες, ε, δουλεύουν για λογαριασμό άλλων, είχαν λιγότερες παραγγελίες. Έτσι δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν υποσχέσεις. Υποσχέσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της ε, διάσκεψης κορυφής του G8 στην Τοβίλ στη Γαλλία. Υποσχέσεις από πλευράς των ανεπτυγμένων χωρών ε, ότι θα βοηθούσαν τις ε, χώρες της Αραβικής Άνοιξης. Μάλιστα είχαν μιλήσει για 8 με 10 δις δολάρια ως βοήθεια στην οικονομία της χώρας μου, ώστε η Τινησία να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πολλά ε, επίμονα αιτήματα των νέων ανέργων κυρίως. Ωστόσο, δυστυχώς, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε συγκεκριμένα. Αυτά τα δέκα δις δολάρια που υποσχέθηκαν στις, ε, στους Τινήσιους δεν δόθηκαν. Και επίσης διερωτώμεθα, αυτά τα δις γιατί δεν δόθηκαν, λόγω του αποτελέσματος των εκλογών ή η ευρωπαϊκή κρίση ευθύνεται για την ε, αθέτηση των υποσχέσεων. Εγώ πραγματικά διερωτώ και είναι θεμητή, θεμητό αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις. Πάντως δεν ήρθαμε σήμερα εδώ να ζητήσουμε βοήθεια, ούτε για να ζητήσουμε να τηρηθούν οι υποσχέσεις που έγιναν τότε, που δόθηκαν τότε. Ε, είχαμε, ήρθαμε για να πούμε πως ε, και, ε, η να σας πω ότι η Αμερικανική οικονομία ωφελήθηκε πάρα πολύ από τη βοήθεια που έδωσε στην Ευρώπη μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και η βοήθεια, και αυτό, αυτή η στήριξη ήταν αμφίδρομη. Η, Ευρώπη στήριξε την, με τη σειρά της την Πορτογαλία και την Ισπανία όταν αυτές ε, επανήλθαν στη δημοκρατία μετά από κάποια χρόνια. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση ωφελήθηκε από την στήριξη που προσέφερε προς την Ανατολική Ευρώπη. Ολόκληρη η Ευρώπη ωφελείται από την οικονομική ανάπτυξη που γνωρίζει αυτή τη στιγμή η Ανατολική Ευρώπη και με τον ίδιο τρόπο ζητάμε και εμείς να γίνουν επενδύσεις επενδύσει κανείς στις χώρες Αραβικής Άνοιξης σημαίνει εμπιστοσύνη στο μέλλον. Είναι επενδύσεις ε, μέσο και μάκρο αλλά πιστεύω πως κάτι τέτοιο θα είναι προς όφελος όλων. Ε, και όλα αυτά βέβαια για τις χώρες που αναπτύσσονται δημοκρατικά. Θα είναι προς και των δύο μερών. Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Υπάρχει πραγματικά αισιοδοξία. Υπάρχει κάποιο όραμα για το μέλλον. Υπάρχει εμπιστοσύνη στο μέλλον για να επενδύσουμε στις, για να γίνουν επενδύσεις στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης. Και όταν λέω ε, Αραβική Άνοιξη, ε, συμπεριλαμβάνω και το Μαρόκο σε, αυτήν, σε αυτές τις χώρες, ακόμα και αν εκεί δεν έγινε επανάσταση, γιατί η Αραβική Άνοιξη είναι η άνοιξη της δημοκρατίας και πιστεύω πως τα αδέρφια μας του Μαρόκου ε, ακολούθησαν αυτό το κίνημα, ακόμα και αν το ακολούθησαν από διαφορετικό δρόμο. Νομίζω πως ο χρόνος που μου είχατε δώσει εξαντλήθηκε. Αυτά ήθελα ωστόσο να τονίσω και μια τελευταία σημαντική παρατήρηση. Τα οικονομικά μέτρα ε, σύμφωνα με την Ισλαμική <laughs> θεωρία. Στην οι οικονομικές αυτές αρχές ισλαμικές ε, βρίσκονται στην οικονομία την ισλαμική και μάλιστα το Λονδίνο και το Παρίσι και η Νέα Υόρκη προηγήθηκαν. Εμείς ε, θαρρύναμε τις ισλαμικές τράπεζες και μάλιστα έχουμε μείνει πολύ πίσω αν συγκριθούμε με τις ε, ευρωπαϊκές χώρες. Και αν δημιουργηθεί ένα ταμείο, αυτό ε, θα μοιάζει με την ε, γαλλική καθολική βοήθεια, για παράδειγμα. Είναι ενώσεις, σύνδεσμοι που βοηθούν τους στοχούς. Και αυτό δεν έχει να κάνει με Ισλαμική ιδεολογία, αλλά με τις ανάγκες των λαϊκών και φτωχών στρωμάτων που χρειάζονται βοήθεια. Δεν πιστεύω πως υπάρχει καμιά Ισλαμική θεωρία που να είναι αντίθετη οικονομικά με τις αρχές του διεθνούς εμπορίου ή του ΠΟΕ. Αντιθέτως, η Ισλαμική οικονομία είναι φιλελεύθερη και ενθαρρύνει την ε, προσωπική ατομική πρωτοβουλία και στον τομέα αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε και κανένας φόβος. Ότι δηλαδή θα μπορούσαν να υπάρχουν ισλαμικές θεωρίες που θα ήταν αντίθετες με τις διεθνείς οικονομικές θεωρίες. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας έδωσα και δύο λεπτάκια επιπλέον, αλλά εν γέννη μείνατε στο χρόνο που σας έδωσα και τώρα θα δώσω το λόγο στον ε, δόκτορα Σαμέχα Φαουζή Χέναν Σας ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το Ίδρυμα Κάρνιτζι που μας κάλεσε εδώ. Και νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία να συζητήσουμε την οικονομική κατάσταση, της θρησκευτικής ελευθερίας, τα δικαιώματα των πολιτών και την δόμηση του νέου κράτους στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης. Θα προσπαθήσω να διευρύνω λίγο το πεδίο εφαρμογής, να μιλήσουμε λίγο πιο ευρέως για την πολιτική οικονομία στην Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένης ε, και της πτυχής των αμυγός οικονομικών ζητημάτων. Καταρχάς, η Αιγυπτιακή οικονομία ακόμα πλήττεται από μια σημαντική ύφεση και η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες συσσωρεύονται αναφορικά με την ε, ανάκαμψη της οικονομίας, ε, την ε, αξιοπιστία της αγοράς, την θεσμική ανασφάλεια, μια αντίληψη αστάθειας, η οποία και αυτή εξακολουθεί να επηρεάζει με αρνητικό τρόπο την οικονομική ανάπτυξη στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τη κυβέρνηση. περιμένουμε 2% μόνο ανάπτυξη φέτο Και στο νέο οικονομικό έτος 2013-2014, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομίας, στο συνέδριο Σούρα, να αναφέρω επίσης ότι τα ποσοστά ανεργίας κινούνται γύρω στο 13% και ο μέσος, η μέση διάρκεια η μέση διάρκεια ενεργείας είναι τρία έτη για το 40% των ανέργων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι πιο πολλοί άνεργοι είναι τα άτομα που μόλις έχουν ολοκληρώσει την ε, εκπαίδευση, την εκπαίδευσή τους. Η νέα γενιά η οποία καλεί και ζητά ελευθερία και δικαιοσύνη στην Αίγυπτο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την αγανάκτησή τους, τον φόβο τους, το θυμό τους για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε έναν νέο προπολογισμό 820 εκατομμυρίων σε ό,τι αφορά δηλαδή ε, επενδύσεις ε, επιπλέον 200 εκατομμύρια Αιγυπτιακές λίρες. σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής, σε ό,τι αφορά τα τέλη για υπηρεσίες ε, γρήγορου διαδικτύου. Κοιτώντα λοιπόν πώ έχει τρέχουσα κατάσταση. Τα τεράστια προβλήματα με τα οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Προκειμένου να σταθεροποιήσουμε την οικονομία, να καταπολεμήσουμε την διαφθορά, να υπάρξει καθολική ανάπτυξη. Διαπιστώνω ότι η κατάσταση λοιπόν είναι πολύ περίπλοκη, πολύ πολύ σύνθετη και ανησυχητική. Η μακροοικονομική σταθεροποίηση προαπαιτεί εφαρμογή μη δημοφιλών πολιτικών σε μια χώρα όπως η Αιγυπτός. Αυτό τι σημαίνει μείωση των ε, επιδοτήσεων, αύξηση της φορολογίας και τέτοιες πολιτικές θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε κοινωνικές αλλά και πολιτικές αναταραχές. Αν η κυβέρνηση προσπαθήσει να επιβάλλει τέτοια νέα μέτρα χωρίς να υπάρχει μια ευρία συνένεση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών φορέων συμπεριλαμβανομένης και της αντιπολίτευσης ειδικά, θα προκαλέσει μεγαλύτερη πολιτική αστάθεια. Και αν η κυβέρνηση από την άλλη προσπαθήσει να αναβάλει την εφαρμογή τέτοιων μέτρων, δίνοντας ε, εξαιρετική οικονομική αρρωγή μπορεί ενδεχομένως να αναβάλει την επίλυση του προβλήματος, αλλά αν θα σκάσει τελικά η κατάσταση θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Άρα, για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τα μέτρα αυτά στο κοινό, θα πρέπει να οικοδομηθεί πρώτα πολιτική συνένεση μεταξύ των πολιτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων κυρίως των ομάδων της αντιπολιτεύσης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς συζήτηση. Χωρίς τη συζήτηση μάλιστα πολύ δύσκολων θεμάτων σε ό,τι αφορά το εκλογικό δίκαιο, την ε, αναθεώρηση του συντάγματος, την μεταρρύθμιση του δικαστικού. Κάποια θέματα τα οποία είναι φλέγοντα στην παρούσα φάση σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αν θέλουμε να σταθεροποιηθεί λοιπόν η πολιτική κατάσταση, η Αίγυπτος θα πρέπει να προβεί σε συμβιβασμούς. Αν θέλει να οικοδομήσει ένα πιο σταθερό δημοκρατικό σύστημα στην Αίγυπτο. Έχω κάποια καταλητικά σχόλια. Αναφέρθηκα στο σύνολο της κατάστασης, στα στατιστικά στοιχεία τα οποία διατίθενται σε αυτά που προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, στον ανταγωνισμό που υπάρχει σήμερα μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης. Κάποια καταλητικά σχόλια, επιτρέψτε μου. στα οποία έχω καταλήξει μετά από έρευνες και ως ε, στο, στο Κοινοβούλιο, αλλά και σε ό,τι αφορά επιστημονικές έρευνες. Καταρχάς, χρειάζεται ένα ευρύτερο όραμα ανάπτυξης στην Αίγυπτο σήμερα και αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση σήμερα. Αν θέλουμε να υπερβούμε τα τρέχοντα οικονομικά προβλήματα, θα πρέπει αναπόφευκτα να επανέλθουμε στα σλόγγαν της Επανάστασης. Κοινωνική πολιτική ελευθερία και όλα αυτά τι σημαίνουν ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα όραμα ανάπτυξη που θα περιλαμβάνει διάφορα τμήματα τη κοινωνία τη Αιγύπτου και με βασικό στόχο πάντα την πρόοδο. Δυστυχώ, ω τώρα δεν υπάρχει κοινωνικό όραμα. Ή, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν το έχω διακρίνει πουθενά. Κοιτώντα τι συζητήσει που διεξάγονται σε διάφορα μέσα ενημέρωση, διαπιστώνουμε ότι οι πιο πολλέ συζητήσει επικεντρώνονται στα θέματα διαφθορά σε διαμάχες μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, αλλά πουθενά δεν βλέπω καμία φιλόδοξη ιδέα σε ό,τι αφορά την πρόοδο της εκπαίδευσης, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση μιας πραγματικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην, Ευρώπη, στην Αίγυπτο. Αυτό που θράβα το είδα. Επίσης ε, διακρίνω ένα αυταρχικό ύφο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. στην Ήπετρο βασικό καθήκον είναι να εμπλακεί ο κόσμος στην οικοδόμηση ενός κοινωνικού κεφαλαίου προκειμένου να υπάρξει τελικά και η οικονομική ανάπτυξη. Με ανησυχία, επίσης το, τα ποσοστά φτώχειας στην Αίγυπτο. 25% στις πόλεις και 50% στην Βόρεια Αίγυπτο. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε λοιπόν την φτώχεια γιατί η φτώχεια προκαλεί πολλά προβλήματα, βία, θρησκευτικέ εντάσεις και πολλά άλλα. Και μπορεί να προκαλέσει επίσης πολλά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια χωρίς ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης. Δεύτερο σχόλιο. δεν είμαι σίγουρος ότι η τρέχουσα κυβέρνηση μπορεί να πετύχει πραγματική οικονομική αναδιάφρωση και αλλαγή σε μια χώρα όπως η Αίγυπτος. Δεν πιστεύω ότι η πολιτική στάση της τρέχουσας κυβέρνησης είναι υπεύθυνη. Θεωρώ ότι είναι μάλλον αδύναμη, ανίκανη να επικοινωνήσει με μεγάλα τμήματα του Αιγυπτιακού λαού. Δεν τίθεται θέμα ανταγωνισμού μεταξύ Ισλαμιστών και λαϊκών δυνάμεων. Πολλές ε, Ισλαμικές ε, δυνάμεις ε, καλούν, απευθύνουν τα βέλη της κριτικής τους κατά της κυβέρνησης και καλούν να αλλάξει η κυβέρνηση. Δεν είναι ικανοποιημένοι με την απόδοση της κυβέρνησης σήμερα. Κατά τρίτον, τρίτο επικριτικό σχόλιο, αν θέλετε, δεν μπορώ να διαχωρίσω τα κοινωνικονομικά ε, δικαιώματα από τα αμυγός τεχνικά δικαιώματα. Ένα παράδειγμα να σας δώσω από την πρωινή συζήτηση και παραθέτω σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τις σχετικές ελευθερίες στην Αίγυπτο. Μπορώ να πω ότι κάποιες από τις κριτικές εντάσεις προκύπτουν από κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Επίσης όμως διαπιστώνω ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση κάποιων τμήματων του Αιγυπτιακού λαού και κατά των χριστιανών. Αυτό σε διάφορες περιστάσεις διαπιστώνεται. Αλλά αν ο κόσμος ε, αποφασίσει για παράδειγμα να μεταναστεύσει και είναι ε, πραγματικά ανησυχητικό το φαινόμενο αυτό. Κάποιοι χριστιανοί αποφασίζουν να μετανεύσουν. Άτομα με καλές συνδέσεις αποφασίζουν να φύγουν και έτσι έχουμε μια διαφυγή αν θέλετε εγκεφάλων από την Αίγυπτο. Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ υψηλότερα στην χριστιανική κοινότητα. Χάνουμε λοιπόν ανθρώπινο κεφάλαιο, κοινωνικό κεφάλαιο και φυσικά οικονομικό κεφάλαιο. Τέλος, να αναφερθώ σε αυτά που είπε η Πρόεδρος για την Ισλαμική θεωρία της οικονομίας. Εξ όσων ε, καταλαβαίνω και το παρακολουθώ το θέμα αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον, δεν έχω δει όμως ως τώρα να υπάρχει κάποια πλήρη οικονομική θεωρία Ισλαμική για την οικονομία στα βιβλία, αλλά στην πράξη τα Ισλαμικά κόμματα όταν έχουν την εξουσία ε, περιμένουν από αυτά να έχουν ε, κοινωνικές πολιτικές που να απεικονίζουν, να αποτυπώνουν το Ισλαμικό δόγμα. Δεν βλέπω να υπάρχει οποιαδήποτε αντίφαση μεταξύ των ε, Ισλαμιστών να αναφερθώ στο θέμα των δανείων, το οποίο είναι καυτό ζήτημα στα πλαίσια του Συμβουλίου Σουρέ. Στην Ανοβουλή. Τίφεται λοιπόν θέμα θρησκευτικής ε, άδειας, θρησκευτικής ελευθερίας Επιλεξιμότητα για δάνεια μεταξύ των διαφορών κομμάτων της Άνω Έχει έρθει ο καιρός να παραμερίσουμε τις φιλοσοφίες, τα θεωρητικά δόγματα. Έχει έρθει ο καιρός να επικεντρωθούμε σε πολιτικές που θα ωφελήσουν τον λαό. Αν έχουμε δημοσιονομικές πολιτικές που θα αποτυπώνουν τις βασικές αξίες του Ισλάμ, θεωρώ ότι αυτό θα δώσει μια καλή ορμή για να σημειωθεί μια αλλαγή στην κοινωνία μας. Αλλά θεωρώ ότι ως τώρα οι πολιτικές που έχουν προταθεί αποτυπώνουν μάλλον νεοφιλελεύθερες τάσεις στην οικονομία, χωρίς να γίνεται κάποια διάκριση λόγω της θρησκευτική, αν θέλετε, διάστασης. Περιμένουμε ακόμα. Μήπως και δούμε να αναπτυχθεί στον τομέα των οικονομικών μια Ισλαμική πολιτική, η οποία θα αποτυπώνει μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή που ακολουθείτε ως τώρα, η οποία, πρέπει να σας πω, δεν έχει αλλάξει καθόλου από το καθεστώς του Μουμπάρακ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Δόκτωρ Χένεν. Τώρα θα δώσω το λόγο στην δόκτωρα Χακίμα Φάσλη, που είναι η επόμενη μας καλεσμένη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ. Στο όνομα του ελεήμονος και μεγαλόψυχου Θεού, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι εδώ και ευχαριστώ εκ βάθου καρδία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση που μου επίθυνε για τη συμμετοχή μου στην διάσκεψη αυτή που στόχο έχει ε, να αντιληφθούμε καλύτερα τι συνέβη στην Αραβική Άνοιξη μακριά από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις για να μπορέσουμε έτσι να αντιληφθούμε όλοι τι συνέβη στην περίοδο αυτή τι συμβαίνει τώρα και να ευοδοθούν και να τελεσφορήσουν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ του αραβικού κόσμου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2009 οι αραβικές χώρες ε, βίωσαν μια σημαντική αλλαγή που χαρακτηρίστηκε ως Αραβική Άνοιξη. Ήταν πραγματικά μια περίοδος ε, διαφωτισμού δύσκολου, αλλά διαφωτισμού και μετάβασης προς μια πιο δημοκρατική και πιο σύγχρονη χώρα από κάθε άποψη, οικονομική, πολιτική, κοινωνική. Και μάλιστα το Μαρόκο ε, δεν έμεινε στο περιθώριο αυτής της διαδικασίας. Οι Μαροκινοί ε, αφομοίωσαν την Αραβική Άνοιξη με πολύ μεγάλη ευφία και από το μονάρχη μέχρι τον απλό πολίτη όλοι οι Μαροκινοί πολίτες συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα το οικονομικό, το κοινωνικό και το πολιτιστικό. Ανοίγοντας διάπλατα τις θύρες ε, σε μια νέα σύγχρονη χώρα που θα είναι όμως πιστή στη, στον πολιτισμό της, στην παράδοσή της και στις διεθνείς δεσμεύσεις της και στραμμένη προς το μέλλον. Το 2011 ήταν μια πολύ πλούσια σε αλλαγές χρονιά. Το πρώτο τρίμηνο του 10 δημιουργήθηκε μια δυναμική κατάσταση που είχε ως αποκορύφωμά της την ομιλία του βασιλέως και τις εκλογές που, που έβγαλαν μια νέα κυβέρνηση και έδωσαν την νίκη στην, στο κόμμα της ελευθερίας και δικαιοσύνης που ανέλαβε για πρώτη φορά τα ενία της εξουσίας. Ευελπιστούμε ότι η νέα αυτή κυβέρνηση θα ανταποκριθεί στις ελπίδες και τις ανάγκες του Μαροκινού λαού και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή και για, το, για τη χώρα και διεθνώς με πολλές χώρες έχουμε ε, διμερείς συμφωνίες, ε, έχουμε και την ε, συμφωνία εταιρική σχέσης, αλλά και ταυτόχρονα βιώνουμε ακόμη τους μετασυσμούς από την Αραβική Άνοιξη. Έχουμε πολλές ε, προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Έχουμε μια μεσαία τάξη που έχει πληγεί, ταλανίζεται από την δύσκολη οικονομική κρίση, αλλά είναι και ο κρογωνιαίος λίγο η ραχοκοκαλά της κοινωνίας. Είχαμε και μία ε, μέγαλο αστική τάξη, μία ελίτ που ε, έγινε πιο πλούσια και μία μικροαστική τάξη που έγινε πιο φτωχή, κάτι που μεγάλωσε το κενό μεταξύ των δύο τμήματων της κοινωνίας. Επίσης, ε, έχουμε και πολλούς νέους που αποκτούν ένα επίπεδο ανώτατης μόρφωσης. Όπως έλεγα λοιπόν, αυτή η τάξη, η κοινωνική τάξη των νέων πλήττεται από μία αφόρητη και σοβαρή ανεργία. Χρειάζονται κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει, αλλά ακόμη δεν έχουμε δρέψει τους καρπούς αυτής της μεταρρύθμισης εξαιτίας της διαφθοράς, της ε, άδικης κατανομής του πλούτου, της φοροδιαφυγής, της απάτης και της κοινωνικής αδικίας. Η κυβέρνηση υπέβαλε ένα νέο πρόγραμμα με κάποιες προτεραιότητες που ενέκρινε η Βουλή. Για παράδειγμα, να επικεντρωθούμε στη διαμόρφωση μιας ε, σύγχρονης χώρας, να δώσουμε νέο δυναμισμό στις αραβοαφρικανικές σχέσεις και να, από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είμαστε σημαντικά. Για παράδειγμα, να ενισχύσει και να κινητοποιήσει κάποια ταμεία για τους απόρους, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, και να ε, βελτιώσει την παιδεία με κατάλληλη χρηματοδότηση. Μάλιστα, η κυβέρνηση δημιούργησε 50.000 νέες θέσεις εργασίας στα πλαίσια του νόμου για τα οικονομικά για το 2012-2013. Επίσης ε, εγκαινιάστηκαν ε, πολλά σημαντικά έργα υποδομής που οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να, ε, να εφαρμόσουν. Επίσης ενισχύσαμε και το Ταμείο Αποζημιώσεων ξεκινήσαμε μια φορολογική μεταρρύθμιση. Η κυβέρνηση της χώρας μου συζήτησε εκτενώς το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης. Μια άλλη μεταρρύθμιση αφορά την αναθεώρηση του νόμου του 1990 για την οικονομική αναδιοργάνωση. Ε, η σε αυτή τα καρπό συνεργασία της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση. Μάλιστα ξεκινήσαμε και τη μεταρρυθμίση των συνταξιδοτικών ταμείων. Ξεκινήσαμε έναν το αγώνα κατά της διαφθοράς. Μεταρρυθμίσαμε τους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες και δημόσιες συμβάσεις. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια διαφανή διακυβέρνηση. Σε γενικές γραμμές λοιπόν η παρούσα κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει και το κόμμα μου προτιμά την μεταρρύθμιση με σταθερότητα όμως και με επιδίωξη της δημοκρατικής διαδικασίας. Στηριζόμαστε στην εθνική ενότητα και στο άνοιγμα. Διαφυλάσσοντας όμως την ε, ε, κοινωνική, περιφερειακή και μουσουλμανική μας ταυτότητα. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Τώρα, καθώς ο στόχος είναι να προχωρήσουμε σε ανταλλαγή όσο, απόψεων όσο γίνεται πιο ανοιχτή, θα δώσω το λόγο σε δύο μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας που το ζήτησαν και μετά σε δύο μέλη Αιγύπτους. Ε, από το ακροατήριο. θα σας ζητήσω να περιορίσετε τις ερωτήσεις σας γιατί πρέπει να ακούσουμε και την ε, εισηγήτρια μετά. Σε δύο λεπτά λοιπόν θα περιορίσετε τις ομιλίες σας και θα είμαι πολύ αυστηρή. Okay, thank you very much. I will be very brief. Uh, thank you for interesting presentations. I would like to ask the... Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Ντρόμπα. Θέλω να ε, ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Αιγύπτου ποια είναι τα σχεδιαζόμενα μέτρα για να χειριστούν το πληθυσμό γιατί ξέρουμε πως η, Αιγύπ... η Αίγυπτος έχει τετραπλασιάσει το πληθυσμό της από το 1907 Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 85 εκατομμύρια κόσμος, πράγμα το οποίο προκαλεί και πολλά προβλήματα. Ε, ποια είναι τα μεσοπρόθεσμα σας οικονομικά σχέδια και μέτρα για να μπορέσετε να χειριστείτε όλον αυτόν τον πληθυσμό, τον απίστευτο που έχετε. Και δεύτερον, ε, η διαφορά ανάμεσα στα Ισλαμικά κόμματα τα οποία ε, δημόσια στηρίζουν το πρότυπο κοινωνικής κατανομής, θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε και σοσιαλιστικό μοντέλο απέναντι στη βασική ισλαμιστική προσέγγιση ε, προς την οικονομία που φαίνεται να είναι φιλελεύθερη και προσανατολισμένη στην αγορά. Ξέρω πως υπάρχουν προβλήματα με τα επιτόκια, ήδη το αναφέρατε, πως αυτό είναι κατά της θρησκείας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, να αντιμετωπίσουμε σε και την ε, πραγματικότητα του σημερινού τραπεζικού κόσμου. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να το χειριστείτε αυτό το θέμα. Uh, Αυτή η ερώτηση βασικά απευθυνόταν στον ομιλητή, στους ομιλητές από την Αίγυπτο. Οπότε, σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε ή προτιμάτε στο τέλος. Επόμενη ερώτηση από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ. Ο Υπουργό κ. Μπεν Σαλάμ αναφέρθηκε στο σχέδιο Μάρσαλ που εφαρμόστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μίλησε για κάποιες αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη και τις ε, μεταβάσεις και τις πολιτικές και τις δημοκρατικές. Δυστυχώς ε, στην Ανατολική Ευρώπη δεν δεχτήκαμε τόσο δαψιλή βοήθεια όπως το σχέδιο Marshall, όπως αυτό, όπως έλαβε η Δυτική Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έγιναν βέβαια κάποιες επενδύσεις ε, με την αλλαγή της κατάστασης και επενδύσεις έγιναν και στην Ουγγαρία, όπως είναι λογικό και φυσιολογικό. Στην αρχή έγιναν κάποιες επενδύσεις ε, που εξυπηρετούσαν και τις δύο πλευρές και στην Ουγγαρία και αλλού και μετά τις αλλαγές της Αραβικής Άνοιξης εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για επενδύσεις και στις αραβικές χώρες. Ε, δηλαδή θα θέλαμε και στη, στον αραβικό κόσμο να δημιουργηθεί ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον και μια οικονομική βάση που θα επιτρέπει την ανάπτυξη. Στην Ουγγαρία έχουμε πλούσια γεωργία και αυτό μας βοήθησε πολύ. Και κάτι άλλο. Αναφέρθηκε το Ισλαμικό πρότυπο τράπεζας. Δεν είναι μόνο θρησκευτικό το ζήτημα, γιατί ξέρω ότι η, η Ισλαμική θρησκεία απαγορεύει την εισπράξη τόκων ε, για τη χορήγηση δανείων. Πώς πιστεύετε θα εφαρμοστεί αυτό στην σύγχρονη εποχή. Μάλιστα. Θέλει άλλος κανείς από το ακροατήριο το λόγο ε, ή κάποιος ευρωβουλευτής να θέσουν ομιλίες. Ωραία, συγγνώμη. Όχι, τώρα δεν το λόγο στον καλεσμένο μας από την Αίγυπτο. Και ο Τελευταίος κύριος που ζήτησε το λόγο, παρακαλώ, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Θα κάνω ένα σχόλιο που απευθύνεται και στους δύο καλεσμένους. Έχω κάποια έγγραφα του Υπουργείου Βιομηχανίας. Θέλουμε να αναπτύξουμε τον ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν θα καταφέρουμε να αναπτύξουμε την εθνική βιομηχανία αν δεν ε, επιλύσουμε τα προβλήματα και του δημόσιου τομέα. Γιατί εκεί έγιναν κάποιες ιδιωτικοποίησεις χωρίς να αποζημιωθούν ε, οι εργαζόμενοι που έχασαν τη δουλειά τους ε, και βρέθηκαν ξαφνικά στο δρόμο. Αν θέλουμε να είμαστε Ανταγωνιστική και στο μέλλον, θα πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις μας ε, τον επόμενο χρόνο. Έχουμε μετά την Επανάσταση αποκαταστήσει κάπως ε, το επίπεδο της παραγωγής μας και πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη μεταπητική βιομηχανία αλλά και στον τομέα των υπηρεσιών Επίσης να αναμίξουμε τους επιχειρηματίες και τους βιομηχάνους ε, στη χάραξη των πολιτικών αλλά και στην εφαρμογή τους. Κάποιος αναφέρθηκε στον νόμο που ισχύει για την κοινωνία των πολιτών. Βρίσκεται σε πολύ προκαταρκτικό στάδιο ακόμη η χάραξη, ο σχεδιασμός αυτού του νομοσχεδίου και υπάρχουν διάφορες τάσεις. Μία τάση ε, εσωστρέφειας ε, με πολύ περιορισμό και χωρίς κανένα άνοιγμα. Δεύτερη τάση που είναι υπερβολικά ανοιχτή, χωρίς όμως καμία διασφάλιση. Και μια τρίτη τάση μιλάει για άνοιγμα προς την κοινωνία, ε, την εξωτερική και την κοινωνία των πολιτών, αλλά και με κάποια χέγγια για την πράσπιση της εθνικής ασφάλειας. Και μάλιστα κάποιες ενώσεις και οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω χρηματοδότησης περισσότερο. Πολύ συχνά οι τοπικές οργανώσεις παραβιάζουν την νομοθεσία για την ε, χρηματοδότησή τους και την ε, ε χορήγηση δωρεών. Εγώ μελέτησα την αντίστοιχη νομοθεσία των ΗΠΑ και του ΗΠΑ και βλέπω ότι εκεί είναι πολύ πιο δρακόντια τα μέτρα από αυτά που θα περιλαμβάνει το δικό μας νομοσχέδιο για τις οργανώσεις και ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να σας πω ότι ο κατάλογος των ομιλητών έχει κλείσει πλέον, γιατί αν ε, τον αφήσουμε ανοιχτό δεν θα καταφέρουμε να μιλήσουν όλοι. Και δεν θα καταφέρουν να απαντήσουν και οι πανελίστες και ούτε καν ο εισηγητή. Να περάσουμε στον επόμενο μιλητή, ο κύριος Μπαρακάτ από το Βελγίο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον Υπουργό Σαλέμ. Μιλήσατε για την βοήθεια που υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάμαι μια μικρή ιστορία τη στιγμή που γινόταν ε, η διάσκεψη της Ντοβίλ. Οι τίτλοι των αραβικών εφημερίδων ήταν «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ υπόσχονται 550 ε, δις ε, δολάρια για να βοηθήσουν τις νέες νεογέννητες δημοκρατίες στον αραβικό κόσμο» και κάτω-κάτω στην ίδια σελίδα υπήρχε η εξή είδηση «Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεδριάζει στις Ριξέλλες για να βρει 10 δις δολάρια για να σώσει την Ελλάδα» δύσκολα τα βρήκαν αυτά τα δέκα δις. Απευθύνομαι λοιπόν στους Ευρωπαίους συμπολίτες μου. Όταν απευθύνεστε στον αραβικό πληθυσμό, προσπαθήστε λιγάκι να είστε πιο συγκεκριμένοι. Δεν θα έλεγα να είστε έντιμοι, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην δίνετε φρούδες ελπίδες, γιατί ο κόσμος ε, πιάνεται από κάποιες ιδέες. Προσβλέπουν στην Ευρώπη, βλέπουν την Ευρώπη ως ε, χώρα ε, δωρητή και όταν οι υποσχέσεις αυτές δεν υλοποιούνται, επικρατεί μεγάλη απογοήτευση. Δεύτερο σημείο, κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για το χρηματιστήριο του Παρισιού, το Λονδίνο Λονδίνου, της, ε, το Βρυξελών ως η Ισλαμική οικονομία. Εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν τους ενδιαφέρει η δομή της ε, Ισλαμικής οικονομίας. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να συγκεντρώσουν, να ελκύσουν ε, τα δις που έχουν οι Ισλαμικές τράπεζες, κυρίως στις χώρες του κόλπου. Δεν τους ενδιαφέρει το ίδιο το σύστημα. Ε, επίσης, όσον αφορά την οικονομία την Ισλαμική, αν αυτή η Ισλαμική οικονομία την οποία υπόσχονται τα Ισλαμικά κόμματα που έχουν πάρει την εξουσία βασίζεται στον ε, φιλελευθερισμό που έχει αποδείξει την αποτυχία του και που έχει φέρει την Ευρώπη και δεν μιλώ για κανονικό φιλελευθερισμό αλλά για τον άγριο φιλελευθερισμό ε, και αποδεικνύει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή ιδρύματα Μα οδήγησαν τι Ευρω... χώρε αραβικές να συμμετέχουμε σε αυτόν τον φιλε... άκρατο φιλελευθερισμό, πιστεύω πω είναι πλέον ο καιρό οι αραβικέ χώρε να βρουν άλλα συστήματα, ανταλλαγέ μεταξύ τους, ε, νοτο σε αραβικέ χώρε για να κάνουν οικονομία. Και ένα αστείο να σα πω, ναι, ναι, ολοκλήρων. Διακόπτη, πρόεδρε. Εντάξει, θα σα το πω μετά, με συγχωρείτε, θα σα πω το αστείο αργότερα. Επίσης ευγενικά να σας πω ότι έχετε κάνει σχόλια που είναι δικαίωμά σας αλλά δεν θέσατε καμία ερώτηση. Περνώ στον επόμενο μιλητή που είναι ο κύριος Μαρζούκ και έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ έχετε δύο λεπτά όπως και οι υπόλοιποι. Θα ήθελα να απευθύνω τα σχολιά μου στον κύριο Φάουση. Δεν θα πρέπει να είναι απόλυτα αρνητική η εικόνα που δίνουμε για την Αίγυπτο και την κατάσταση που επικρατεί στην Αίγυπτο. Έχουμε και άλλα οικονομικά νέα, γιατί μπορέσαμε να να κτίσουμε κάποια κονδύλια τα οποία είχαν φύγει από τη χώρα μας. Πρόκειται για χρήματα, δυο λομελιτέα ποσά και έχει υπάρξει πρόοδος και όσον αφορά τη γεωργία, ιδιαίτερα το στάρι. Αυτό που θα θέλαμε λοιπόν είναι να, υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις. Εμείς δεν ζητάμε βοήθεια, ε, περισσότερες επενδύσεις ζητάμε. Και ο κύριος Μοχάμπετ Μπεν είχε πει πως αυτές οι επενδύσεις θα είναι προς όφελος όλων και συνέκρινα την κατάσταση με τα ωφέλη τα οποία αποκόμισαν οι ΙΠΑ από το σχέδιο Μάρσαλ. Όσον αφορά την ε, αντιπολίτευση του κόμματος, ε, τις θέσεις μάλλον του κόμματος Νουρ. Οι θέσεις μας δεν βασίζονται στη θρησκεία, αλλά έχουμε ένα οικονομικό όραμα το οποίο έχουμε υποβάλει στο κοινοβούλιο και ο κύριος ε, Σαμέχ είναι μέλος του κοινοβουλίου αυτού χρειάζονται πιστώσεις ε, και δάνεια ε, για να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία μας. Δεν θα πρέπει δηλαδή όλα αυτά να τα δούμε μόνο από, το οπτικό, από την οπτική γωνία της θρησκείας. Ευχαριστώ. Μπραμ, from the Netherlands. Εγώ έχει κύριε Μπραμ από την τώρα. Έχετε δύο λεπτά. Ναι, δεν θα χρειαστώ καν δύο λεπτά. Καταρχάς, μια πρώτη ερώτηση στον κύριο Ανίν και στον Υπουργό Μπεντσάλεμ. Η περιφερειακή οικονομική συνεργασία είναι αρκετά περιορισμένη στην περιοχή τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Ποιε θεωρείτε λοιπόν ότι είναι οι προοπτικέ για περαιτέρω περιφερειακή ολοκλήρωση και έχετε την αίσθηση ότι οι οικονομίε τη περιοχή είναι συμπληρωματικέ αρκετά προκειμένου να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα ενοποιημένο σύνολο. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και εμείς στην Ολλανδία προασπιζόμαστε, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια κινητήριο δύναμη για την οικονομία στις, ε, στην περιφέρεια αυτή. Πώς θα μπορούσατε να προσπαθήσουμε λοιπόν να πείσουμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διστάζουν σε ό,τι αφορά μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα για θέματα αγροτικών προϊόντων, λέει η Πρόεδρος. Μετά από αυτά, λοιπόν, να δώσω το λόγο για Ζήκη. Um, where, <laughs> Okay. Εδώ είμαι, Πρόεδρε. Η ερώτησή μου έχει να κάνει, είναι προς τον ε, Υπουργό Γεωργίας, κ. Μπενσάλεμ, να πω ότι μου προκάλεσε κάποια έκπληξη η έλλειψη οικονομικού ράματος από την Τινησιακή κυβέρνηση αλλά και από τις άλλες κυβερνήσεις από τα Ισλαμικά νέα κόμματα. Είναι σαν να μην έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει τις τελευταίες, τα τελευταία χρόνια. Οι επαναστάσεις που έχουν ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές ρίζες. Και φαίνεται ότι ξεχνάμε ότι η τελευταία δεκαετία ήταν δεκαετία οικονομικής ανάπτυξης. Αίγυπτος νομίζω ότι είχε 5% ανάπτυξη ένα έτος ε, και την Ισία νομίζω και η Συρία και παρά την ανάπτυξη αυτή αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα με την ενεργία των νέων. Πού είναι λοιπόν οι πολιτικές, πού είναι τα οράματα, η δημοσιονομική, η χρηματοοικονομική πολιτική, η εμπορική πολιτική. Δεν βλέπουμε τίποτε άλλο, μόνο την Ισλαμική, τα Ισλαμικά οικονομικά, την Ισλαμική οικονομική πολιτική. Μιλάτε για ένα καθεστώς ε, ευεργεσίας, όχι για οικονομία ουσιαστικά. Πώς μπορούν λοιπόν τα Ισλαμικά κόμματα να δημιουργήσουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που χρειάζονται στις, στην κάθε χώρα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, ο κ. Ουλγκέν. My question is with Έχω μία ερώτηση για το μέλλον της Αιγυπτιακής οικονομίας και θα ήθελα να μου πει τη γνώμη του Δ. Χάινεν. Όταν βλέπουμε σήμερα την Αίγυπτο, νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε ότι είναι άθλια οικονομική κατάσταση, τεράστια ανεργία, μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα δύσκολη οικονομική συγκυρία. Φαίνεται να πλησιάζει το χείλο της οικονομικής καταστροφής αν δεν γίνει τίποτα για να, για αναταχθεί αυτή η κατάσταση. Και όταν βλέπουμε τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις σε άλλα αναπτυσσόμενα κράτη, διαπιστώνουμε ότι η οικονομική κρίση ουσιαστικά πυροδότησε την έναρξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. Όπως λένε, θα πρέπει να πηγαίνει χαμένη μια καλή κρίση στα θέματα της οικονομικής μεταρρύθμισης. Αλλά ούτε και αυτό είναι σίγουρο. Σε άλλες περιπτώσεις η οικονομική κρίση ε, ενίσχυσε την πολιτική αστάθεια ή την, επέ, την ε, επιδίνωσε περαιτέρω την κατάσταση. Στο Αιγυπτιακό πλαίσιο πώς α, λειτουργεί η κρίση. Βλέπετε, καταρχήν αντιλαμβάνεστε την οικονομική αιγυπτιακο πλαισιο πως λειτουργει η κριση πιστεύετε να θα κατάληξε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αν ε, ζήσετε κι εσείς οικονομική κρίση. Θεωρείτε ότι θα φέρει αυτό του εταίρους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ώστε από κοινού να ε, χαράξουν το μέλλον της χώρας ή θεωρείτε ότι θα επιτείνει μια τέτοια οικονομική κρίση την πολιτική αστάθεια και θα ενισχύσει τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση. Τελευταίος ομιλητής τώρα, ο κύριος Νόρμαν. Okay. Σας ευχαριστώ. Έχω δύο παρατηρήσεις και δύο ερωτήσεις και θα προσπαθήσω αυτό να τα υποβάλω σε δύο λεπτά. Συμφωνώ με τον κύριο Μπερσάλεν ότι συνεχίζεται η άνοιξη στην Τινησία. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο για το μέλλον, πολύ συγκρατημένα για την ακρίβεια. Δεύτερη παρατήρηση για το σχέδιο Μάρσαλ για τις υποσχέσεις που δεν ε, τηρήθηκαν. Όντως, ε, και διαρωτόμαστε πού οφειλόταν αυτό. Το Ταμείο ή Ταμείων ε, υπήρχε έλλειψη προθυμίας και βούλησης από την παρούσα κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε περισσότερο επενδύσεις παρά τέτοια βοήθεια. Και δύο ερωτήσεις. Λυπούμε, αλλά διαφωνώ για το ότι δημιουργήθηκαν 132.000 θέσεις εργασίας. Γιατί βλέπουμε, αν ήταν τόσες πολλές, θα βλέπουμε τον αντικτυπό τους στην ε, την οικονομία. 100.000 άνθρωποι μπορεί να μπήκαν στο δημόσιο τομέα, στο δημόσιο στην Τινησία, κάτι που επιβάρυνε ουσιαστικά τον, το δημόσιο της Τινησίας. Έχουμε 85% του προϋπολογισμού που χρηματοδοτεί το δημόσιο και η αιτήσια αύξηση του προϋπολογισμού αυτού είναι 7%. Απλούστατη ερώτηση λοιπόν. Πώς θα μειώσετε αυτό το 85% ε, για να ανατάξουμε κάπω την οικονομία μα. Γιατί αλλιώ μέσα σε δύο χρόνια θα χρεοκοπήσουμε. Αν ένα τόσο μεγάλο τμήμα του προπολογισμού αφιερώνεται στη χρηματοδότηση του δημοσίου και των δημοσίων υπαλλήλων, τη δημόσια διοίκηση. Επίσης, ε, δεν θα πρέπει η ανάπτυξη να γίνεται από φιλαθροπικέ κοινωνικέ οργανώσει, παρόλο που έχουν πολιτικό προσανατολισμό. Πότε, πώς θα μειώσουμε έτσι ε, τον κίνδυνο να χρησιμοποιούνται δημόσια κονδύλια για να προβάλλονται κάποιες πολιτικές οργανώσεις απλώς. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Ε, ήταν πολύ χρήσιμη η συμβολή σας και η συμμετοχή σας στη συζήτηση. Πολύ εύστοχα τα σχόλιά σας και σημαντικές ερωτήσεις. Πολλές ερωτήσεις ε, αφορούσαν την Αίγυπτο. Φοβάμαι λοιπόν ότι θα δυσκολέψουν τον Αιγύπτιο καλεσμένο μας. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να ξεκινήσω από εσά, κύριε Έινεν, ή θέλετε λίγο περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστείτε. θα ξεκινήσετε εσείς, πολύ ωραία. Και έχετε πέντε ολόκληρα λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και για τις ερωτήσεις σας. Αυτό σημαίνει ότι ε, οι πιο πολλοί από εσάς θεωρείτε την Αίγυπτο ακρογωνιαίο λίθο στην ε, περιοχή και πρέπει να σας ε, απαντήσω συνοπτικά σε, σε κάποια από τα πιο βασικά ερωτήματα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη δημογραφική πολιτική. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζει κάτι τέτοιο στην ε, Αίγυπτο. Καταλαβαίνετε, τα δημογραφικά προβλήματα είναι πολύ πιεστικά για χώρες που θέλουν να πετύχουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Αλλά δυστυχώς οι πιο πολλές από τις κοινωνικές πολιτικές της Αιγύπτου μετά την Επανάσταση ουσιαστικά έχουν υπονομευθεί, έχουν επισκιαστεί. Γιατί η κοινωνία πιο πολύ επικεντρώθηκε σε αμυγός πολιτικά ζητήματα, σε Νομίζω ότι τα συμβούλια τα οποία κληρονομήσαμε από το παλιό καθεστώς ε, θέλουν να υπάρχει μια δήλωση της αποστολής τους. Δηλαδή η κοινωνία θέλει καταρχάς φυσικά σταθερότητα, να συζητιούνται κοινωνικές πολιτικές, γιατί βλέπουμε αντικρουόμενες τάσεις στην Αίγυπτο σήμερα. Κάποιοι λένε ότι έχουν σημειωθεί επιτεύγματα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και ότι αυτά αποτελούν κληροδότημα του παλιού καθεστώτος. Έτσι το εκλαμβάνουν ορισμένοι. Άλλοι πάλι λένε ότι πρόκειται για ένα κληροδότημα της ίδιας της κοινωνίας. Και ότι προσπιζόμαστε τα δικαιώματα των γυναικών και αυτό αποτελεί καρπό των προσπαθειών της ε, κοινωνίας μας και δεν θα έπρεπε να αποδίδονται τα εύσημα στο παλιό καθεστώς για το θέμα αυτό. Οι κοινωνικέ πολιτικέ λοιπόν έχουν κάπω παραμεριστεί και θα πρέπει να επικεντρωθούμε πιο πολύ σε αυτέ. Δυστυχώ όμω. Αυτό δεν συμβαίνει. Το δεύτερο ζήτημα σε ό,τι αφορά την Ισλαμική θεωρία και τα... την οικονομική πολιτική. Έχουμε μια Ισλαμική κυβέρνηση, δεν θέλω να μιλήσω εξ ονοματό τη, αλλά να σας πω ποια είναι η προσωπική μου άποψη. Τα Ισλαμικά κινήματα συμπεριλαμβάνουν μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Ε, τη μέση τάξη, πλούσιους ανθρώπους, ε, εργάτες, όλους τους περιλαμβάνουν. Στην Ισλαμική κοινωνία και κοινότητα υπάρχουν πολιτικές ε, αντιλήψεις πολύ διαφορετικές. Ως πολιτικός όμως και ως ε, ε ακαδημαϊκός εστιάζομαι πιο πολύ στις ε, πολιτικές που συζητιούνται στην Αναβουλή, που συζητιούνται στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Δεν θέλω να επικεντρωθώ σε θέματα ιδεολογικά, αλλά θέλω να επικεντρωθούμε στην πολιτική που αφορά τα καθημερινά κοινωνικά πολιτικά προβλήματα και ως τώρα δεν ε, διαφαίνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην επίλυση και την αντιμετώπιση των καθημερινών μας προβλημάτων. Σίγουρα. Ο συνάδελφος από το Κοινοβούλιο ανέφερε κάποια επιτεύγματα. Ναι, προφανώς. Κάθε μέρα κάτι καινούργιο παράγουμε. Και κάποια υπουργεία λειτουργούν σωστά και καλά στην ε, Αίγυπτο. Όταν μιλώ όμως για την κυβέρνηση, μιλώ για ένα ενιαίο πολιτικό σώμα με συγκεκριμένη ευθύνη. Δεν μιλώ μονομενα, για μεμονωμένα επιτεύγματα. Μιλώ για το σύνολο. Τα συνολικά επιτεύγματα της κυβέρνησης. Και δεν είμαι ικανοποιημένο με τα συνολικά επιτεύγματα Τη κυβέρνηση και νομίζω ότι πολλέ πολιτικέ ομάδε, πολλοί πολιτικά κόμματα και πολλοί πολιτικοί στην Αίγυπτο ασκούν κριτική, έντονη κριτική. Ακόμα και το κόμμα της ε, ελευθερίας και της δικαιοσύνης ασκεί έντονη κριτική ενάντια στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν πρέπει ανοιχτά να το δηλώσουμε. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα, ένα βασικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο τώρα, νομίζω ότι είναι ανταγωνιστικές οι οικονομίες του αραβικού κόσμου. Το μεγαλύτερο τμήμα των προβλημάτων είναι πολιτικής φύσεως. Μιλώντας ε, με τους Άραβες, θα ήθελαν ασφαλώς όλοι οι Άραβες ε, να συνενωθούν. Αλλά υπάρχουν πολλά πολιτικά εμπόδια και ελπίζω το πνεύμα της Αραβικής Άνοιξης να μας συνενώσει πιο πολύ. Και όταν συνενωθούμε οικονομικά, θεωρώ ότι θα ακολουθήσει και πολιτική ένωση. Γιατί ξέρετε, η οικονομία είναι πάρα πολύ ισχυρή και μπορεί πραγματικά να ενώσει τους λαούς. Τέλος. Και αν δεν έχω ξεχάσει καμία ερώτηση, να αναφέρω ένα ζήτημα το οποίο θα ήθελα να διευκρινιστεί και να μην υπάρχουν πλάνες σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα σε καιρούς πολιτικής μετάβασης προς ένα δημοκρατικό καθεστώς, θα ήθελα να αναφερθώ στον Φίλιπ Σιμίτα, ο οποίος μελέτησε τις εμπειρίες που προκύπτουν από τις νεοναδιόμενες δημοκρατίες σε παγκόσμιο επίπεδο σε περιόδους μεταβατικές είναι πολύ πιο σωστό να επαφείται κανείς σε ικανές κυβερνήσεις που μπορούν να πετύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και να βελτιώσουν την κοινωνία και να θέσουν, αν θέλετε, την κοινωνία στο σωστό δρόμο. Αυτό εννοώ όταν μιλώ για μια ικανή κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε ικανή κυβέρνηση η οποία να παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα, να δώσει την αίσθηση στον λαό ότι πραγματικά υπάρχει διαφορά. Αυτό αφενός. Αφετέρου, θα ήθελα να αναφέρω επίσης τον Φράνσις Φοκουγιάμα, όταν μίλησε για την εμπειρία της Ιαπωνίας μετά τον πόλεμο. Ανέβρε ότι η Ιαπωνία δεν χτίστηκε με χρήματα, χτίστηκε από τον κόσμο, από τα άτομα που κατήχαν τις θέσεις κλειδί στον κρατικό μηχανισμό. Αυτοί είχαν το όραμα, εργάστηκαν σκληρά έσπηραν, αν θέλετε, το πνεύμα και τους καρπούς του, της εργασίας στην κοινωνία και στην νεολαία και δημιούργησαν ένα νέο, μια νέα ανατροπία. Αυτό αναζητούμε και θα αποτελέσει ένα βασικό εμπόδιο το οποίο θα κληθούμε να επερπηδήσουμε στην Αίγυπτο. Ίσως και σε άλλες χώρες της Αραβικής Άνοιξης, αλλά δεν θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος άλλων χωρών. Στην Αίγυπτο χρειαζόμαστε όμως τέτοια δυνατότητα διακυβέρνησης μια διακυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία θα δώσει μια καλύτερη αίσθηση στον κόσμο και θα δώσει την αίσθηση στον κόσμο ότι κάτι αλλάζει στην καθημερινή του ζωή. Ευχαριστώ. Very Σας ευχαριστώ. Όντω είχατε πολλές ερωτήσεις, γι' αυτό και σας επέτρεψα να παραβείτε κάπου στο χρόνο σας. I hope that not everybody will do this. Uh, now I give the floor to... Και να δώσω το, τώρα το λόγο στον Υπουργό Μπεν Σαλέμ γιατί πολλές ερωτήσεις απευθυνθήκαν και σε εκείνον. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Όντως είναι μεγάλη πρόκληση να απαντήσει κανείς σε τόσο πολλές ερωτήσεις μέσα σε 5-6 λεπτά, αλλά προσπαθήστε το. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, όταν μίλησα για το σχέδιο Marshall, δεν είπα ότι το σχέδιο Marshall κάλυψε και την Ανατολική Ευρώπη μαζί με τη Δυτική. Εννοούσα ότι η βορειοαμερικανική οικονομία υποφελήθηκε από τις συνέπειες, από τις επιπτώσεις που είχε το σχέδιο Μάρσαλ. Και οι οικονομίες των χωρών της Δυτικής Ευρώπης επωφελήθηκαν από την βοήθεια που χορήγησαν στις χώρες πρώην Ανατολικής Ευρώπης. Είχα μια συνάντηση με τον πρέσβη της χώρας στην Τινησία και μιλήσαμε για κάποια σχέδια γεωργικής ανάπτυξης και προγράμματα άρδευσης. Και επιθυμούμε διακαώς τη συνεργασία με την Ευρώπη, τόσο την Ανατολική όσο και τη Δυτική. Στην Τινησία αυτό που επιθυμούμε είναι όσοι θέλουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε μια παραδοσιακή τράπεζα και να έχουν ένα εισόδημα να μπορούν να το κάνουν. Αλλά όσοι θέλουν να διαλέξουν μια Ισλαμική τράπεζα και αυτοί να έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Υπάρχει δικαίωμα επιλογής, κάτι που στο παρελθόν δεν ήταν δυνατό. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών για τους πολίτες, ώστε να μπορούν ελεύθερα να διαλέγουν πού θα καταθέτουν τις οικονομίες τους. Και για να απαντήσω στον ε, βουλευτή από το Βέλγιο, θα ήθελα να πω ότι όταν είπα ότι το Ισλάμ ε, τάσεται υπέρ μια φιλελεύθερη οικονομία. Δεν εννοούσα τη ανεξέλεγκτη απελευθέρωση, τον ακρεφνή φιλελευθερισμό, σε καμία περίπτωση. Η Ισλαμική οικονομία είναι μια οικονομία που έχει μια φιλελεύθερη χρειά, αλλά και μια κοινωνική κατεύθυνση. Η Ισλαμική οικονομία σε καμία περίπτωση δεν ε, αντιβαίνει στις ε, αρχές ε, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Ο Ευρωβουλευτής από την Ολλανδία μίλησε για την περιφερειακή συνεργασία και είπε ότι η περιφερειακή συνεργασία δεν ε, αξιοποιήθηκε δεόντως. Δυστυχώς είναι αλήθεια αυτό εξαιτία των δικτατορικών καθεστώτων, γιατί οι δικτάτορες είχαν πολύ συγκεκριμένα ατομικά συμφέροντα. Και όταν ο Μπεναλή θύμωνε με τον Καντάφη, έκλεινε τα σύνορα για ολόκληρους μήνες. Θέλουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Και είμαστε υπέρ της περιφερειακής εργασίας, όχι μόνο με τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης, αλλά γενικώ με τις χώρες της περιοχής. Όπως σας είπα όμως υπάρχουν ακόμη περιφερειακά προβλήματα, όπως το πρόβλημα της Σαχάρας, που παρεμποδίζει τη δημιουργία ενός, ε, μιας περιφερειακής ενότητας, την ε, ούμα δηλαδή, την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ. Θέλουμε μια συνεργασία που βρίσκει σύμφωνος και τους λαούς της περιοχής. Ε, σε αυτήν προσβλέπουν, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια περιφερειακή συνεργασία. Αλλά υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο οχθών της Μεσογείου, της Βόρειας και της Νότιας. Κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερος. Ε, επίσης δεν είπα ότι... Α, δεν συμφωνώ με την διαπίστωση ότι η Αίγυπτος δεν έχει οικονομικό όραμα. Δυστυχώς μέσα σε ένα πεντάλεπτο δεν μπορούσα να δώσω λεπτομέρειες. Αυτό οφειλόταν έλλειψη χρόνου όμως, όχι σε έλλειψη οράματος, γιατί πραγματικά το Ισλαμικό Οικονομικό Πρόγραμμα είναι εξαιρετικά πλούσιο και ενδελεχές. Αν μου δίνει λίγο χρόνο η Πρόεδρος, θα σας πω ότι το προηγούμενο οικονομικό μοντέλο στηριζόταν σε ανάπτυξη μόνο των παράκτιων περιοχών. Οι παράκτιες περιοχές θεωρούνταν η ατμομηχανή της οικονομίας, ενώ οι υπόλοιπε περιοχές ήταν απλά βαγόνια του σειρμού. Το 84% των επενδύσεων πήγαιναν στις παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ η υπόλοιπη ε, χώρα, που ήταν και πολύ πιο φτωχή, λάβανε το υπόλοιπο 16% που ήταν και αμεληταίο σε σχέση με το 84% που πήγαινε στις παραθαλάσσιες ζώνες. Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας επενδυόταν, το 76% του προπολογισμού αυτού επενδυόταν στην ενδοχώρα. Σε 14 δηλαδή από τις 24 συνολικά επαρχίες. Στο παρελθόν είχαμε ατμομηχανή στο βορρά, την παραθαλάσσια ζώνη και οι υπόλοιπε επαρχίες ήταν τα βαγόνια του σειρμού. Εμείς τώρα θέλουμε να αντιστρέψουμε αυτή την τάση, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ενδοχώρα και να γίνει κάθε βαγόνι από μόνο το ατμομηχανή, αν μου επιτρέπετε αυτόν τον παραλληλισμό, το σιδηροδρομικό. Και τώρα έχουμε πιο πολλέ ατμομηχανέ και όχι μόνο μία. Ο κύριο Μανφέρη, που είναι φίλο τη Τινησία, είπε ότι δεν συμφωνεί ότι δημιουργήθηκαν 230.000 θέσει εργασία. Εγώ δεν είπα 230.000, είπα ότι δημιουργήθηκαν 132.000 θέσει εργασία. Πάντως μπορεί να διαφωνούμε στην ανάλυση, αλλά θα πρέπει πάντα να συμφωνούμε στους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί είναι ουδέτεροι, δεν είναι θέμα ανάλυσης. Πρόκειται για αριθμητικά στοιχεία που μας δίνει η ανώτατη στατιστική υπηρεσία. Δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος λοιπόν στους αριθμούς. Αν κάναμε τέτοια λάθη θα μας ξεμπρόσχεζαν μέσα σε δύο λεπτά στο facebook. Εμείς έχουμε τα στοιχεία αυτά από την Εθνική Στατιστική μας Υπηρεσία και κανένας δεν τα αφισβητεί. Έχουμε 20.000 θέσεις εργασίας από το 2012 που ουσιαστικά όμως άρχισαν να λειτουργούν από το 2013. Σε ό,τι αφορά τι θέσει εργασία στη δημόσια διοίκηση, θα ήθελα να σα δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Μέσα σε πέντε χρόνια στο Υπουργείο Γεωργία συνταξιοδοτήθηκαν 5.800 υπάλληλοι και προσλήφθηκαν μόνο 760. Οπότε η τιμησιακή διοίκηση, δημόσια διοίκηση, παρόλο που έχει υπαλλήλου, ε, δεν θεωρούμε ότι έχει αρκετούς υπαλλήλου. Χρειαζόμαστε προσλήψεις μερικές φορές βαθμό για να στελεχώσουμε το Υπουργείο Γεωργίας μας. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που πρέπει να είμαι αυστηρή και να σας κόβω το λόγο, αλλά δυστυχώς δεν έχω άλλη επιλογή, γιατί διαφορετικά θα... δεν θα προλάβω να μιλήσουν όλοι όσοι πρέπει ακόμα να μιλήσουν. Δόκτωρα Αφάσλη, σας δίνω το λόγο με τα χαράς. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ πιο σύντομη από ό,τι προηγουμένω, ε, αν και δεν μου απευθύνθηκε κάποια ερώτηση, ωστόσο είναι μια ευκαιρία. Ίσως αυτό γιατί ήμουν πολύ σαφής. Έχω τρία, ε, τρία πράγματα που θέλω να αποσαφηνίσω. Το ένα είναι μια ερώτηση που έθεσε σήμερα το πρωί ένας βουλευτής που είπε ότι δεν κατάλαβε πώς μπορούμε να πούμε ότι το, το κοινωνικό κίνημα ε, στο Μαρόκο είναι ένα κίνημα κατά ε, της πείνας. Το κίνημα αυτό η, περιπτώσει, η Αραβική Άνοιξη που γνώρισε το Μαρόκο ήταν ένα κίνημα υπέρ της αξιοπρέπειας, ίσως να ήταν ένα πρόβλημα μετάφρασης. Δεν μιλάμε για πείνα, αλλά για αξιοπρέπεια. Ε, δεύτερη παρατήρηση, πιστεύω πως η σημερινή μας συνεδρίαση είχε στόχο να μιλήσει για το αντίκτυπο των Ισλαμικών κομμάτων στην οικονομία. Στο Μαρόκο εμείς επιλέξαμε την αλλαγή στο πλαίσιο της σταθερότητας και αυτό ε, θέλετε ενσωματώνει μια συμμετοχική προσέγγιση γιατί κατά τη γνώμη μας ένα πολιτικό κόμμα που έχει Ισλαμική αναφορά καταρχήν είναι πολιτικό κόμμα η Ισλαμική αναφορά είναι μια αναφορά που καθορίζει κατά κάποιο τρόπο Συγκεκριμένε ενέργειε ή διαβήματα, αλλά, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα πάντα και ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να, βελτιω... να δει πώ θα βελτιώσει τον τρόπο ζωή τι συνθήκε διαβίωση των πολιτών. Ένα σωρό καινούργια πράγματα έγιναν από τη νέα κυβέρνηση του Μαρόκου. Πριν από λίγο μίλησα για το Ταμείο Αποζημιώσεων και ένα σωρό άλλε μεταρρυθμίσει. Αυτή τη στιγμή γίνονται τέτοιε μεταρρυθμίσει, ώστε κάθε υπουργό αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει κάποιο κεφάλαιο μεταρρυθμίσεων, ούτως ώστε να φτιαχτεί έτσι μια νέα δημοκρατία και για να σας πω και μια ιστορία, το νέο σύνταγμα έχει επιφέρει μια νέα καινοτομία, υποχρέωση δηλαδή του αρχηγού κυβερνήσεων να έρχεται μια φορά το χρόνο για να μιλήσει για τα οικονομικά προβλήματα. Σήμερα η ακροματικότητα που της συζήτησης των επικεφαλής ε, της κυβέρνησης ε, ε, ήταν πολύ ψηλότερη από την ακροαματικότητα των τελευταίων ποδοσφαιρικών αγώνων. Μπάρσα Μπάγερν, φανταστείτε. Και αυτό το λόγο για να σας καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή έχω έχει συμφιλειωθεί ο απλός πολίτης με την πολιτική και σε τέτοιο βαθμό που πλέον όλοι μιλούν για την πολιτική, όλοι συζητούν για το τι κατάφερε ή δεν κατάφερε η κυβέρνηση. Στο Μαρόκο δηλαδή προσπαθούμε, όπως σας είπα, να εγκαθιδρύσουμε αυτήν την προσέγγιση του δικαιώματος στη διαφορά του δικαιώματος να έχει κανείς διαφορετική άποψη. Ζητώ συγγνώμη, απασπιπτώ είμαι αρκετά σύντομη. Ναι, ναι, δεν υπάρχει λόγος να ζητάτε συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και έτσι φτάνουμε στο τελευταίο τμήμα αυτού του πάνελ που είναι πολύ σημαντικό γιατί πρόκειται για την σύνοψη που περιμένουμε από την εισηγήτριά μας, την κυρία Σάρα Σάγιες. Σας ευχαριστώ πολύ. Να προσπαθήσω, αντί να επαναλάβω αυτά που είπαν όλοι, να προσπαθήσω να εξαγάγω αυτά που θεωρώ ότι ήταν τα πιο βασικά συμπεράσματα, τα πιο βασικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να σκεφτούμε στο μέλλον. Νομίζω ότι ο κύριος Χάναν ξεκίνησε λέγοντας, ε, μιλώντας για πολιτική οικονομία. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο αναδύθηκε από το πάνελ αυτό. Δεν μπορούμε να αμελήσουμε τις πολιτικές διαστάσεις των οικονομικών συνθήκων στις ανερχόμενες αυτές χώρες και να τις διαχωρίσουμε από τέτοια θέματα. Πραγματικά δεν έχει νόημα. Υπάρχει λοιπόν μια εσωτερική και μια εξωτερική πτυχή. Η εσωτερική πτυχή, όπως είπε η κυρία Σφάσλη, πώς κατανέμεται η ανάπτυξη. Δεν επαρκεί ιδιαίτερα σε αυτές τις χώρες να μιλάμε για ανάπτυξη, ΑΕΠ, και τέτοιους όρους, τέτοια στατιστικά στοιχεία, τα οποία δεν αποτυπώνουν ουσιαστικά το πώς ο κόσμος βιώνει την οικονομία. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πολιτικό και οικονομικό ζήτημα, να δούμε πώς κατανέμεται ε, η ανάπτυξη στον κόσμο. Και ένα βασικό στοιχείο που οδήγησε στις επαναστάσεις ήταν η ιδιοκτησία, αν θέλετε, του πλούτου που άνοιγε ουσιαστικά σε ένα πάρα πολύ μικρό τμήμα του πληθυσμού και αυτό προκαλούσε στρεβλώσεις στην οικονομία με ένα έντονο συνέστημα αδικίας, το οποίο οδήγησε σε πολιτική έκρηξη. Άρα θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιο είναι ο ρόλος των νέων ε, κυβερνητικών κομμάτων, των Ισλαμικών κυβερνητικών κομμάτων, γιατί αυτό αποτελεί και το θέμα του συνεδρίου, αλλά και το ρόλο όλων των κομμάτων σε ό,τι αφορά ε, τη λογοδοσία για τα εγκλήματα, τα οικονομικά του παρελθόντος και τον αντίκτυπο που είχαν στον κόσμο προκειμένου να μην συνεχιστούν στο μέλλον αυτές οι πρακτικές, γιατί η σταθερότητα των νέων κυβερνήσεων εξαρτάται όχι μόνο από την ικανότητά τους να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και το καθεξής, αλλά και από το κατά πόσον θα διορθώσουν αυτό το αίσθημα, το βαθύ αίσθημα αδικίας που επικρατεί ένα αμυγός πολιτικό ζήτημα. Ο κύριος Χάναν μίλησε για την ε, πολιτική συνένεση η οποία προαπαιτείται για να περάσουν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται είτε από εξωτερικού παράγοντε είτε από εσωτερικού οικονομικού παράγοντε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί η οικονομική συνένεση ουσιαστικά παρεμποδίζεται από πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ε, θρησκεία, με την κοινωνία, με όλα τα ζητήματα που συζήτησαμε και σήμερα το πρωί. Με την ελευθεροτυπία, με του δημοσιογράφου. Αυτή η πολιτική συνένεση λοιπόν δεν υπάρχει. Αντιθέτως, πώς μπορεί κανείς να περάσει τις βαθιές οικονομικές τομές που απαιτούνται. Επίσης, ε, τέθηκε το θέμα της οικονομικής χρηματοδότησης, ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά τις οργανώσεις που ασχολούνται με ανθρωπιστικό έργο. Αυτό είναι ένα ευρύ ζήτημα το οποίο μας απασχολεί όλους και στις δυτικές οικονομίες και δημοκρατίες. Το ζήτημα του ποιος είναι ο αντίκτυπος των τεράστιων ε, αξιώσεων, των τεράστιων απαιτήσεων σε χρήμα, προκειμένου να ασκηθεί πολιτική. Και αυτό επηρεάζει και την οικονομική πολιτική, γιατί όταν η πολιτική οικονομική ε, καθοδηγείται από πολιτικά συμφέροντα, αυτό περιορίζει και τις οικονομικές πολιτικές που μπορεί να εφαρμοστούν. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο τέθηκε προς το τέλος είχε να κάνει με την ε, προθυμία του ανθρωπίνου κεφαλαίου να συμμετάσχει στην ανάπτυξη νέων οικονομικών πολιτικών βάσει της πολιτικής τους ε, πεποίθησης. Ανάλογα με το ποιο ε, έχει την εξουσία. Δηλαδή ότι ο κόσμος σε πολλέ περιπτώσει δεν συμμετέχει στη δικασία αυτή επειδή δεν εμπιστεύεται τα κόμματα που είναι στην κυβέρνηση. Η εξωτερική διάσταση, η πολιτική διάσταση των οικονομικών έχουν να κάνουν με το τι έγινε στις επαναστάσεις σε σύγκριση με την επανάσταση του 89, με το τι έγινε μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, με το τι έγινε με τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και μιλάω ως Αμερικανή. Ανέκυψαν λοιπόν τέτοια ερωτήματα. Γιατί είναι τόσο αδύναμη η εξωτερική αυτή βοήθεια η οικονομική κρίση που επικρατεί σε όλο τον κόσμο, αν θέλετε μία ανασφάλεια σε ό,τι αφορά ε, το πώς διαμορφώνονται αυτές οι κυβερνήσεις μετά την Επανάσταση και επίσης είναι ερωτηματικό για τις πολιτικές αξίες και για το κατά πόσον η οικονομική βοήθεια μπορεί σε, σε, κατά κάποιο τρόπο να συνδεθεί με το σεβασμό κάποιων πολιτικών αξιών σε αυτές τις χώρες μετά την μεταβατική αυτή φάση. Άρα, συγκρίνοντας και πάλι την κατάσταση με την Ευρώπη και την Ιαπωνία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι κάπως άδικη αυτή η σύγκριση. Γιατί η οικονομική αρρωγή χορηγήθηκε με κάποιους συγκεκριμένους όρους, με κάποια εγγύηση πολιτικών αξιών. Άρα η κατάσταση σήμερα είναι κάπως πιο περίπλοκη από ό,τι ήταν τότε. Επόμενο θέμα. Δύο θέματα έχω να αναφέρω ακόμα. Σε ποιο βαθμό, σε ποια έκταση οι εξωτερικές ε, συνθήκες, οι εξωτερικοί όροι που τίθενται σε ό,τι αφορά τη βοήθεια, είτε είναι δάνεια, είτε είναι επιδοτήσεις, σε ποιο βαθμό λοιπόν έχουν ιδεολογικό προσανατολισμό αυτές ε, οι προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, ε, ο φιλελευθερισμός που συνδέεται σε πολλές περιπτώσεις με, τον, με τη διεθνή βοήθεια, με τη διεθνή οικονομική αρρωγή. Η ιδεολογία των δωρητών, των χωρών δωρητών, των οργανισμών που κάνουν τις δωρεές μας οδηγούν στο επόμενο ερώτημα. Ποιο είναι το οικονομικό όραμα των Ισλαμικών κομμάτων. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Γιατί η επίκρατη μεγάλη διχογνωμία στη ΣΥΠΑ και στην ε, Ευρώπη σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα μέτρα λιτότητας, αν είμαστε υπέρ ή κατά. Σε ποιο βαθμό λοιπόν εμείς που αντιμετωπίζουμε αυτή την εσωτερικό διχασμό σε ό,τι αφορά το οικονομικό μας όραμα, μπορούμε να προαπαιτήσουμε ένα σαφές οικονομικό όραμα από τις αναδυόμενες αυτές οικονομίες. των λεχθέντων. Ο κόσμος στις χώρες αυτές μπορεί να αναρωτιέται σε ποιο βαθμό τα Ισλαμικά κόμματα και το οικονομικό τους όραμα πραγματικά αποσκοπούν στην επίλυση των, των συστημικών προβλημάτων των οικονομιών τους όπως ε, έθεσε ο Δόκτωρ Φάζλι στην παρουσίασή του. Σε ποιο βαθμό λοιπόν τα Ισλαμικά αυτά κόμματα προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ισορροπία, την οικονομική ισορροπία ή σε ποιο βαθμό προσπαθούν να τα συγκαλύψουν ουσιαστικά για να συγκαλύψουν τις επιπτώσεις της ανισορροπίας και να πάρουν το μεγαλύτερο μερίδιο της τούρτας, όπως και τα προηγούμενα καθεστώτα. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Εμείς σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε το πάνελ μας. Ως καλή συγγήτρια δώσατε τόσες απαντήσεις όσες ε, και ερωτήσεις κάνατε στη συνέχεια. Έτσι μας δώσατε πολύ μεγαλύτερη τρόφη προς συζήτηση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Έντουαρτ Μακμίλαν Σκότ, για τα καταληκτικά σχόλια. Και μάλιστα σας δίνουμε το χρόνο και δύο λεπτά νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Ευχαριστώ πολύ, Ανέμι. Αυτό είναι προ τιμήν τη εξαιρετική σα προεδρία το γεγονό δηλαδή ότι είμαστε εντό του χρόνου. Εγώ εδώ αντιπροσωπεύω τον πρόεδρο Σούλτ του Ευρωκοινοβουλίου που δεν μπορεί να είναι παρόν. Μου ζήτησε ω αντιπρόεδρο ε, για, υπεύθυνο για αρμόδιο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τι υπερατλαντικέ σχέσει, καθώ και επειδή πολλά χρόνια ε, εγώ ασχολούμαι με την ανάπτυξη και τη μεταρρύθμιση του αραβικού κόσμου και μάλιστα Είχα το προνόμιο να είμαι ο πρώτος εξωτερικός πολιτικός που, που επισκέφθηκε την Αίγυπτο κατά την Επανάσταση πριν από δύο χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν από αυτέ μου τι ιδιότητε να σα ευχαριστήσω όλου που ήρθατε εδώ, να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Κάρνικη, το Ινστιτούτο Edmond, τον Πρόεδρο και του συζητητέ που, που κατέστησαν δυνατή την υλοποίηση αυτή τη διάσκεψη. Η ευρωπαϊκή πολιτική, ειδικά προ του γειτονέ μα, θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματική. Αλλά δεν είναι πάντοτε εύκολο να κατανοήσουμε του γειτονέ μα ε, και τι πολιτικέ αυτέ ε, ιδιαίτερα για του Ευρωπαίου πολίτε. Οι πρωτοβουλίε σαν τη σημερινή διάσκεψη είναι πολύ χρήσιμες γιατί κατασκευάζουν γέφυρες και λειτουργούν υπέρ της κατανόησης για τα όσα συμβαίνουν στην ε, άμεση μας γειτονία και καθώς και μας ε, κάνουν να δούμε το μέλλον κάπως για τη γειτονία. Εγώ ε, θαυμάζω και σέβομαι τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες ξεκίνησαν την Ισία, η Λιβύη και η Αίγυπτος όπως και άλλες χώρες σαν το Μαρόκο στην περιοχή. Η διοργάνωση εκλογών και η σύνταξη ενός συντάγματος είναι πολύπλοκα έργα και εμείς οι Ευρωπαίοι το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό, αλλά θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα από την δικιά μας ευρωπαϊκή εμπειρία. Καταρχήν η δημοκρατία δεν είναι μόνο μια διαδικασία, πρέπει να είναι και αποτελεσματική. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές με 50-1%. Αλλά για να υιοθετήσει σύνταγμα και να σχηματίσει το μέλλον της χώρας χρειάζεται συνένεση πανεθνική και μάλιστα μια υπερπλειοψηφία σε κάποια συστήματα, δηλαδή σχεδόν 75% του πληθυσμού. Πρέπει ο κόσμος να σέβεται τις ιδέες σου και ο καθένας να έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του. Μόνο έτσι μπορούν να φτιαχτούν θεσμικά όργανα τα οποία να αντιπροσωπεύουν το σύνολο του πληθυσμού. Όπως είπε δε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Έλμαρ Μπρόκα, ε, η εναλλαγή αλλά και οι σταθερές ε, ε, αξίες είναι αυτά που χρειάζονται ε, για να λειτουργήσει ένα δημοκρατικό σύστημα. Μια επιλογή, δυνατότητα επιλογής και δυνατότητα α, τον, κανείς να ιτηθεί αλλά και να ξανακερδίσει. Αυτά καθορίζουν τη δημοκρατία. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία όταν δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα, όταν το δικαστικό δηλαδή σώμα δεν είναι ελεύθερο και όταν οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η δημοκρατική διαδικασία και όλοι οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί φορεί θα πρέπει να δείξουν σεβασμό στι δημοκρατικέ αξίε και πρακτικέ. Και αν δεν το καταφέρουμε αυτό, θα είναι το αποτέλεσμα άλλα αυταρχικά καθεστώτα που δεν θα σέβονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των πληθυσμών των χωρών αυτών. Θα πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι έχετε την πλήρη στήριξη του Κοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Όπως ίσως τα γνωρίζετε, το Ευρωκοινοβούλιο κάθε χρόνο τιμά εξαιρετικά άτομα τα οποία έχουν δεσμεύσει τη ζωή τους για τον αγώνα κατά της μη ανοχής, της μυσαλλοδοξίας ε, και το 2011 το βραβείο αυτό δόθηκε σε πέντε ακτιβιστές ε, της Αραβικής Άνοιξης, Αχμέτα Ζουμπαΐντ, Αχμέτα Ζανούση από τη Λιβύη, Ραζάν Ζεϊτούνε και Αλή Φαρζάτ από την Συρία και φυσικά μετά θάνατον και δικαίως τον Μοχάμετ Μποαζίζη της Τινσίας. Ε, αν ξεχνάμε την προέλευσή μας, αν ξεχνάμε ότι οι νέοι, οι γυναίκες, ε, οι, εκείνοι που δεν είχαν δικαιώματα και πάχαζαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, τα, τα, τα ιδρύματα και οι νέοι φρέσκοι θεσμοί θα αποτύχουν. Όταν ο πρόεδρος Μαρζούκη απευθύνθηκε στο Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο φέτος, ε, είπε στην ομιλία του και το υπογραμμίζω ότι αυτές οι επαναστάσεις δεν είναι εθνικιστικές και ξενοφοβικές, αλλά είναι κοινωνικές και και δημοκρατικές. Εμείς ε, θα θέλαμε η καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να γίνει σεβαστή παγκοσμίω και να μην ε, υπόκειται σε θρησκευτικέ ιδιαιτερότητε ή σε ε, άλλες ε, αρχές. Η οικονομική ανάπτυξη είναι κλειδί για τη σταθεροποίηση και πάλι αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει πολύ καλά η Ευρώπη. Δυστυχώς η οικονομική πρόοδος στον αραβικό κόσμο είναι εξαιρετικά αργή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να βρούμε τρόπο να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι και ιδιαίτερα οι νεότερες γενναίε θα έχουν την αξιοπρέπεια, την δουλειά και την ευημερία που πρέπει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σχηματίσουμε ένα ευημερέ και ε, φωτεινό μέλλον για τις χώρες μας. Θα ήθελα να βρούμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε κοινέ προκλήσεις μέσω του αμοιβαίου σεβασμού και της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης και των χωρών σας που πρέπει να αναπτύξουν την ειρήνη και την ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για τη διοργάνωση της σημερινής διάσκεψης και ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές που ήρθαν και συμμετείχαν. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια και για τις σοφές παρατηρήσεις που κάνατε. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης και για να κλείσουμε την διαδικασία αυτή εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο για το αυριανό δε πρόγραμμα που ξεκινά στις 9 το πρωί θα συνεδριάσουμε στα κτίρια του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Rue ε, ε, 1100 Βρυξέλλες δεν είναι πολύ μακριά από εδώ και φυσικά η, η βοηθοί του Ιδρύματος Κάρνεγκη θα σας κατευθύνουν προς το κτίριο αυτό. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, στο πέρας της σημερινής συνεδρίασης, θα έχω τη χαρά να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ, για τις συμβολές σας και να συγχαρώ τους συνδιοργανωτές αυτής της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας ε, συνεδρίας σεμιναρίου που είναι παραπα... ακόμη περισσότερο ενδιαφέρουσα γιατί όπως παρατηρήθηκε επανειλημμένο σήμερα θα είναι, μία από τις... είναι μάλλον μία από τις πρώτες ε, διασκέψεις όπου εκείνοι που προσκλήθηκαν και για τους οποίους τόσο πολλά υπόθηκαν και στους οποίους τόσο σπάνια έχουμε μιλήσει, δηλαδή εκπρόσωποι των κομμάτων που δικαίως ή αδίκως έχουν χαρακτηριστεί ισλαμικά και που παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στις χώρες τους. Για όλα αυτά λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα και καλή δουλειά για αύριο. Ευχαριστώ.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 Lord Balda, βοηθάει και πλάσκο.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 und Herren, die Sitzung ist eröffnet. και κύριοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Περνάμε στην ψηφοφορία για την ε, γνωματότηση της κυρίας Βέιμπερ. Δεν είναι εδώ η κυρία Βέιμπερ και γι' αυτό δεν ε, θα πάρει το λόγο. Περνάμε στην παραγραφό 1. Τροπολογία 1 σε τρία τμήματα. Γκάλερ. Το τμήμα του κυρίου Γκάλερ. Ο οποίος βρίσκεται σε μία αποστολή σήμερα στο Πακιστάν σε μία αποστολή παρατήρησης εκλογών. Δεν είναι και εντελώς ακίνδυνη αυτή η επίσκεψη. Και θα πρέπει να πω ότι υπό τις συνθήκες αυτές ε, το να κάνει κανείς αυτή τη δουλειά θα πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωριστεί. Όταν ε, οι συνάδελφοι έχουν το θάρρος και την τόλμη να κάνουν τέτοια έργο. Κυρία Σχάκη, θέλετε το λόγο, όχι. Α, μάλιστα. Πρόεδρε, συγγνώμη, νόμιζα ότι είχαμε ξεκινήσει την ψηφοφορία. Κύριε Γενική Γραμματέα, ίσως θα μπορούσαμε να το καταγράψουμε αυτό στα πρακτικά ως παράδειγμα. Τώρα, τμήμα 1 της τροπολογίας 1, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρία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 Die Abstimmung ist 48 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση. Θα βρούμε και ποιος αποφάσισε να απόσχει. Περνάμε τώρα στην έκθεση Σχάκε. Έχετε παρατηρήσει ε, συνάδελφε, όχι. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Περνάμε στην 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 59 υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Θεωρώ ότι απορρίπτεται για την 59. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. 25 ψήφι υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές. Να το ελέγξουμε. Θεωρώ όμως ότι και πάλι έχουμε την ίδια πλειοψηφία. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά όμως. Πέρα εφορίας. 30 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Η 62 στην περιορισμένη μορφή υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Και την 65 παρακαλώ. Υπέρ. Για την 65 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Όχι, είδαμε, κάναμε ψηφοφορία δύο φορέ, λέει ο Πρόεδρος. 66, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67, υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται η συνάδελφη Λαντσπέργης με τη βοήθεια των κομμουνιστών, αλλά να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ένα ψηφοφορία. Abstimmung Πέρασε. 24 υπέρ, 28 κατά, δεν απέδωσε η συμμαχία η 68 υπέρ. Κατά. Άποχες. Και αυτή απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το έλεγχο. Έλεγχο για την 74. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. 28 ψήφοι υπέρ, 25 κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην 79 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, εγκρίνεται, συγγνώμη. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές είναι οριακό το αποτέλεσμα. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Για την 83. Πέρας. 26 υπέρ, 29 κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται 90. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 30 ψήφοι υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Άποχες. Η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Ναι, το δέχεστε. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Πέρα ψηφοφορίας. «28 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται». Και συνάδελφος Άριος Βόλσκι ψήφισε τρεις φορές. Αλλά δεν φτάνουν οι ψήφοι. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 101 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ. Είναι οριακό το αποτέλεσμα. Πέρας ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 27 κατά απορρίπτεται. Γιατί είναι 101. 102 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρα ψηφορίας. 26 υπέρ, 29 κατά, απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Για το δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 100... Είχαν ψηφίσει στους σελίστες, λέει ο πρόεδρος. για την 117. Πέρας ψηφορίας. 26 υπέρ, 25 κατά, εγκρίνεται. 116 τώρα. Όχι, 119. Καταπληκτή. Ναι, δίκιο έχετε. 119 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7. Με προφορική τροπολογία. Η εισηγητρία, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να απορρίψω τη συμβαστική, την προφορική τροπολογία και να ψηφίσουμε τη συμβαστική λύση που προέκυψε από τη συνεργασία μας ε, με πολύ επικοδομητικό και συνεργάσιμο πνεύμα. Προτιμώ λοιπόν το κείμενο της συμβαστικής τροπολογίας χωρίς την προφορική. Υπέρ της ε, συμβαστικής 7. Κατά. Έλεγχος. Πέρασα. 30 υπέρ 27 κατά εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στην 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας. 26 υπέρ, 30 κατά, απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Κύριε Σάρισβοσκη, ψηφίζουμε. τη ψηφοφορία. Μας λείπουν ακόμα τρει ψήφοι. 23 υπέρ, 34 κατά, απορρίπτεται. 131 υπέρ. 130, 130 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας ψηφορίας. 27 υπέρ, 32 κατά, απορρίπτεται. 132-136 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 133-137 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στη συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 140 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας. 28 υπέρ, 32 κατά. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά Ήσασταν υπέρ ή κατά, Τζεφρή. Υπέρ. Α, η ψήφο σα ήταν η καθοριστική. Λυπάμαι που το λέω. Εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Άποχες. Και αυτό δεν είναι σαφές. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρασε. 31 ψήφοι υπέρ, 28 κατά, εγκρίνεται. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Έχετε μία ψήφο παραπάνω. Δεν σας χορτάνουμε. 162 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά έλεγχος. Antrag, das ist geschlossen. Πέρα ψηφορίας.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 Κατά. Αποχές έγκρινεται. 171. Στη συνοπτική έκδοση υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Έλεγχος. Έλεγχος για την 171. είσαστε λίγο τεμπέληδες την πρώτη φορά και δεν σηκώσετε τα χέρια σας. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στη συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε την 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Στην 16 περνάμε. Συμβαστική 16, διορθώνει ο πρόεδρος. Συμβαστική 16, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 35, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36. Α, όχι, έχει καταπέσει. 39. Για την 39 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ για τη 40. Πέρας ψηφορία 27 υπέρ, 30 κατά, απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 υπέρ έλεγχος για την 2. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 2. Πέρας ψηφορίας. 33 υπέρ, 27 κατά, εγκρίνεται. Η 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7 και 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος είναι 34 παρακαλώ. Έναρξη ψηφορίας. Πέρας. Τρίαντα υπέρ 27 κατά εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία του συνόλου του κειμένου. Έναρξη ψηφοφορίας. Η τη φορέα. 54 ψήφοι υπέρ, μία ψήφο κατά, μία ψήφο εποχή. Ε, κυρία Μπριζάζοτς, έχετε το λόγο. Επιτέλου. Εκ μέρου του ΕΛΚ θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε πω η έκθεση για την κατάσταση α, στην ελευθεροτυπία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αφορά την κατάσταση στον κόσμο και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να το προσδιορίσω αυτό και να το διευκρινίσω για τα πρακτικά. Ευχαριστώ, θα το συμπεριλάβουμε, αλλά θα ήθελα εκ νέου να υπογραμμίσω το εξή. Ε, καλό είναι να αναφέρεται σε μια τέτοια έκθεση ότι θα πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν αφορά δεν είναι έκθεση για το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δάλλως θα έχουμε προβλήματα με τις άλλες επιτροπές της αρμόδιας, να προσέξουμε θέματα αρμοδιότητας. Γιατί υπάρχει και η σχετική έκθεση από την αρμόδια επιτροπή, γι' αυτό λοιπόν να προσέξουμε. Το πολιτικό ευκταίο το οποίο όμως δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της Επιτροπής ΑΦΕΤ, να μην υπησέλθει υπομορφή τροπολογιών στην ε, Ολομέλεια, να μην κρατεθεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε του κανόνες, του σχετικούς. Αν συμφωνείτε λοιπόν, θα το υποδείξω αυτό και στην υπηρεσία της Ολομέλειας, τη σχετική. Και τώρα περνάμε στην έκθεση μιλανμών.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 Για τη 43 με προφορική τροπολογία. Ρούτσεκ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 46 υπέρ. Όχι. Η 46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην 54. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Και πάλι είναι τροπολογίες που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητα στη ΣΥΝΤΑ. Αλλά θα τις ψηφίσουμε. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 62-63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αλλά ας την ψηφίσουμε, ας την ελέγξουμε. Την 64. Έναρξη πληροφορία. Πέρασα. 23 υπέρ, 33 κατά, απορρίπτεται. Η 65 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε στην 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρινέται και περνάμε τώρα στην συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. Σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα υπέρ. Εγκρίνεται. Α, δεν πείτε μου και ποιοι είστε κατά. Εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα της 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά ας το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφορίας. 23 υπέρ, 34 κατά, απορρίπτεται. 88, λέει ο πρόεδρος.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Στην 39 περνάμε υπέρ, κατά αποχές έλεγχος. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά το ελέγξουμε. Ποιος φώναξε έλεγχο. Πέρας. Ποιος είπε το τσεκ. Ποιος ζήτησε έλεγχο. Εσείς. Κάποιος είπε να το ελέγξουμε. Και τώρα περνάμε στην 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 103. Υπέρ. Κατά αποχές ε, η 103 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 110 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα έχει ρυθμιστεί από μόνο του. Το 111 υπέρ. Α, συγγνώμη. Να ψηφίσουμε και το τρίτο τμήμα της 110 λοιπόν. Υπέρ.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 κατά απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 129. 127 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 136 ως προσθήκη στην 135 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρι... Εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 144. Υπέρ. Κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές σύγκρινεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές έλεγχος πέρας ψηφορίας 25 υπέρ, 33 κατά, απορρίπτεται 170 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 197. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 200 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 202 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 203 έχει καταπέσει 9 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ή 15, ή 15 πρώτα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και περνάμε στην συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 32 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρας ψηφορίας. 26 υπέρ, 30 κατά, απορρίπτεται 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Abstimmung geschlossen. Πέρας 47 ψήφοι υπέρ, 6 ψήφοι κατά, 5 αποχές. Εγκρίνεται. Συνάδελφοι θα ήθελα να κάνω μία πρόταση. Και αν ε, συμφωνείτε να το υποστηρίξετε στις ομάδες σας. Σας παρακαλώ μία στιγμή ησυχία. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Θα ψηφίσουμε τη σύσταση της Επιτροπής ΙΝΤΑ για τις διαπραγματεύσεις ε, το Μάιο. Εμείς ε, θα ψηφίσουμε τον Μάιο, τον Ιούνιο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να τις ψηφίσουμε μαζί τις εκθέσεις αυτές την έκθεση και την γνωμοδότηση. Αν θέλετε λοιπόν να το υποστηρίξετε αυτό στι ομάδε σα για να γίνει μια κοινή συζήτηση το Μάιο, για να μην το συζητάμε δύο φορέ αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά την διαφορετική εταιρική σχέση. Συμφωνείτε παρακαλώ. Θα θέλαμε αυτή η συζήτηση τη διαφορετική σχέση τη Επιτροπή ΑΦΕΤ και τη Επιτροπή Ίντα να συζητηθεί από κοινού. Όχι μία τον Ιούνιο ή άλλη τον Μάιο. Αν θα θέλετε λοιπόν να το μεταβιβάσετε αυτό στις ομάδες σας για να γίνει η σχετική αλλαγή στην ημερήσια διάταξη και θα κάνει η γραμματεία ότι περνάει από το χέρι της για να ρυθμιστούν τα πρακτικά. Ευχαριστώ πολύ και πέρα στη συνεδρία